Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Έχετε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης μπροστά σας. Είστε ικανοποιημένοι όλοι με το σχέδιο ημερήσιας διάταξης, μπορούμε να το εγκρίνουμε. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται λοιπόν η ημερήσια διάταξη. έγκριση τώρα των πρακτικών της συνεδρίασης 24 έως 26 Ιανουαρίου 2011. Μπορούμε να εγκρίνουμε και τα πρακτικά. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και πριν περάσω στο επόμενο σημείο, έχω κάποιες ανακοινώσεις. Μια ανακοίνωση για το σημείο 3. Θα ήθελα να καλωσορίσω μια αντιπροσωπεία του Σουηδικού Κοινοβουλίου από την Επιτροπή Μεταφορών του Σουηδικού Κοινοβουλίου και επισκέπτονται τις Βρυξέλλες και την Επιτροπή μας. Είχαμε ένα πολύ ευχάριστο γεύμα. Σας καλωσορίζουμε. Χαιρόμαστε που είστε εδώ μαζί μας και προσβλέπουμε στη συνεργασία μας και στο μέλλον. Κάθονται όλοι στο πίσω μέρος της αίθουσας. Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε πολύ για την επισκεψή σας. Sorry. Tack. Το επόμενο σημείο, η ανακοίνωση των, της θέσης του Συμβουλίου θα πρέπει να σας ανακοινώσω ότι για τα βαρέα οχήματα και για τη χρήση τους για ορισμένες υποδομές ε, και για τη χρέωση η οποία είναι γνωστή ως ευρωβινιέτα, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ε, ότι σύμφωνα με το άρθρο 61 η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έγκριση της οδηγίας ε, για την χρέωση ε, των βαρέων οχημάτων, ε, θέση η οποία ελήφθη από το Συμβούλιο μαζί με ε, τους λόγους που οδήγησαν στην έγκριση και τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή αυτό σημαίνει, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η περίοδος η οποία υπάρχει τώρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη θέση του σε δεύτερη ανάγνωση αρχίζει από τις 18 Φεβρουαρίου. Αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση του Προέδρου, λοιπόν, για να είναι γνωστό προς όλους. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι οι ψηφοφορίες. Έχουμε πέντε ψηφοφορίες. Αν δεν έχετε την κάρτα σας για την ηλεκτρονική ψηφοφορία, παρακαλώ να μας το πείτε. Εύα, δεν έχεις την κάρτα σου. Βεβαίω, σε σημειώνω να ψηφίσει με του σοσιαλδημοκράτε, σωστά. Όταν φτάσουμε στη ψηφοφορία θα το λέμε κάθε φορά. Θα μας το αναφέρεις κάθε φορά. Κάνε μας ένα σήμα. Λοιπόν, πρώτη ψηφοφορία. Έκθεση Ζασάντα. τροποποιητικό πρωτόκολλο της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ηνωμένων Πολιτειών. Ξεκινάμε με την πρώτη παράγραφο, παράγραφο ε, ε, τροπολογία 3 της κυρίας Λίχτεμπεργκερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 του συγκριτού είναι ίδιο το κείμενο με την τροπολογία Μάισνερ 2. Θα το δούμε μαζί. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Με ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. 22 23 ψήφοι υπέρ, 3 ψήφοι κατά, καμία αποχή εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Ζασάντα. Επόμενο σημείο είναι η πρόταση απόφαση του Συμβουλίου για τη Συμφωνία Αεροπορικών Μεταφορών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Καναδά. Η κυρία Τικάου είναι η συγγήτρια. Δεν έχουμε τροπολογίε. Κατευθείαν την τελική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. 25 ψήφισαν, 27 ψήφι, 27 υπέρ, καμία ψήφος κατά. Συγχαρητήρια, κυρία Τικάου. Το επόμενο σημείο είναι το σημείο του κυρίου Ρικέ, Συμφωνία Ευρωπαϊκών Κοινοτών Βιετνάμ σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών. Τελική ψηφοφορία και άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Πάλι 27 με την ψήφο τη ΕΒΑ. 27 υπέρ, καμία ψήφος κατά. Εγκρίνεται. Επόμενο σημείο. Έκθεση UGS. Απαλλαγή 2009 για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Μία τροπολογία του εισηγητού. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία τώρα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορία. 25 ψήφοι υπέρ, μία ψήφο κατά. Συγχαρητήρια κύριε Ουτζία. Προσθέσαμε και την ψήφο τη κυρία Λίχτεμπέργκερ. Δεύτερη έκθεση του κυρίου Ουτζία. Απαλλαγή 2009 για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Αερομεταφορών. Μία τροπολογία του εισηγητού έχουμε και πάλι Ψήφοι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, αρχιτή ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε η ψηφοφορία. 22 ψήφοι υπέρ, 23 με την κυρία Λίχτεμπεργκερ, 4 ψήφοι κατά, καμία αποχή εγκρίνεται. Και πάλι συγχαρητήρια στον εισηγητή. Το επόμενο σημείο και πάλι στη σειρά των πολλών εκθέσεων του κυρίου Τζίες είναι η απαλλαγή 2009 για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Εδώ έχουμε κάποιες τροπολογίες. Ξεκινάμε τροπολογία 1 Βαντάλλον, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 του εισηγητού, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές να το ελέγξουμε. Για την τροπολογία 5 παρακαλώ να ψηφίσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι, πέρασε τη ψηφοφορία. 12 ψήφοι υπέρ, 14 ψήφοι κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 6 του κ. Βαντάλεν, υπέρ, κατά, αποχές, Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά στο ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 6. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. 16 υπέρ με τη κυρία Λίχτεμπερ και 10 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 7 του κυρίου Βαντάλεμ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. 23 υπέρ, μία ψήφο κατά, τρει αποχέ. Εγκρίνεται. Το επόμενο σημείο, έκθεση Ουτζία και πάλι για την κοινή επιχείρηση ΣΕΖΑΡ, απαλλαγή για το 2009. Μία τροπολογία του εισηγητού και πάλι ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τελική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε 26 υπέρ, μία ψήφος κατά, καμία αποχή, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια για όλες τις εκθέσεις σας, κύριε Ουτζίας, για την απαλλαγή όλων αυτών των οργανισμών. Το επόμενο σημείο είναι το σχέδιο γνωμοδότησης για την απαλλαγή 2009, το Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τμήμα 3, Επιτροπή. Είναι η έκθεση του κυρίου Γκρός, Επιτροπή και Εκτελεστικοί Οργανισμοί. Τροπολογία 1, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές. Να το ελέγξουμε, νομίζω ότι απορρίπτεται. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 1. Εψήφισαν όλοι. Πέραση ψηφοφορία. ψηφοφορίας. 10 υπέρ 16 κατά μία αποχή απορρίπτεται. Για την παράγραφο 4 τώρα έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία από την ομάδα των φιλελευθέρων και μια προφορική τροπολογία για τη δεύτερη γραμμή που αντικαθιστά τη λέξη notes με τη λέξη regrets. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογίες 6 και 7 έχουν αποσυρθεί. Περνάμε λοιπόν στην τελική ψηφοφορία και άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας. Εύα υπέρ. 25 υπέρ, μία ψήφος κατά μία αποχή, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Γκρός. Το, επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης είναι η έκθεση Φιντάντζα για τον τουρισμό στην Ευρώπη. Mr. Fidanza, floor is yours. Κύριε Φιντάντζα, έχετε το λόγο. Grazie, Presidente. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Μετά από αυτή την ανταλλαγή απόψεων ε, στη συνάντηση της Επιτροπής μας ε, στις αρχές του Δεκεμβρίου, τώρα έχουμε μια, είχαμε μια ευρύτερη ανταλλαγή απόψεων με το κείμενο που υποβλήθηκε. Η έκθεση αυτή, όπως το γνωρίζουμε, είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον προσδιορισμό μιας νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τουρισμό βάσει του άρθρου 195 τη συνθήκη της Σαββόνα που προβλέπει τη νέα αυτή αρμοδιότητα για τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την νέα αυτή αρμοδιότητα η Επιτροπή προχώρησε υπό την, με την πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου κ. Ταγιάννη και όποιος δεν παρακολούθησε την υπόθεση να σας υπενθυμίσω ότι η δήλωση της Μαδρίτης του Απριλίου του 2010 τον Ιούνιο του 2010 ακριβώς υπευλήθη το κείμενο της ανακοίνωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 21 δράσεις από την Επιτροπή Ανάπτυξης υπέρ ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τουρισμού και μετά υπό την Βελγική Προεδρία το Συμβούλιο για τον Ανταγωνισμό υιοθέτησε σημαντικά συμπεράσματα που για πρώτη φορά είπαν ότι ο τουρισμός αποτελεί από τις κύριες προτεραιότητες της βιομηχανικής ευρωπαϊκής πολιτικής. Τον Οκτώβριο πέρυσι έγινε αυτό και μετά στο φόρουμ της Μάλτας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα πρώτο σχέδιο για την εφαρμογή αυτής της ανακοίνωσης με τις 21 δράσεις που προβλέπονται. Όπως σας είπα, είχαμε αυτήν την ανταλλαγή υπόψεων αρχές Δεκεμβρίου στην Επιτροπή μας Ταυτόχρονα δε συνεργαστήκαμε με τους κοιόδης εισηγητές σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και ουσιαστικά όλοι συμφώνησαν για τα κύρια σημεία της εργασίας αυτής. Επίσης αποδόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στις απόψεις ε, γνωμοδοτήσεις και άλλων πέντε επιτροπών που εκφράζονται για το κείμενο αυτό σε Επιτροπή ΣΥΙΤΡΕ, περιφερειακή, κουλτούρας κλπ. Και αυτές οι επιτροπές βλέπουμε ότι προχωρούν σε ανακοινώσεις κλπ. σχετικά με το κείμενο αυτό και δύο οι κατευθύνσεις ε, για την εργασία. Να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες και πώς θα εφαρμοστούν πρακτικά αυτές οι 21 δράσεις που προβλέπονται από την Επιτροπή για το σχέδιο εφαρμογή και ταυτόχρονα όμως να δούμε και άλλα στοιχεία τα οποία είναι πέρα από το κείμενο της ανακοίνωσης και εν μέρη πέρα από τις ε, στενές αρμοδιότητες ας πούμε του Αντιπροέδρου Ταγιάννη αλλά είναι ουσιαστική σημασία ε, για να είναι ανταγωνιστικός ο τουρισμός μας. Ε, και σε λίγο, στη σύντομη παρέμβασή μου, θα προσπαθήσω να αναφέρω μερικά από αυτά τα πράγματα. Η Ευρώπη είναι ο τίτλος ε, της εργασίας της Επιτροπής σαν πρώτο προορισμό τουριστικό στον κόσμο και εμείς θέλουμε να εργαστούμε πάνω σε δύο κατευθυντήριες γραμμές. Πρώτα απ' όλα, τι γίνεται, πώς θα ε, ελκύσουμε καλύτερα περισσότερο με, ε, από τις αναδυόμενες αγορές επίσης που δυνητικά υπάρχουν δεκάδες εκατομμύρια νέοι τουρίστες που θα πρέπει να τους προσελκύσουμε στην Ευρώπη να διαλέξουν σαν τελικό προορισμό τους στην Ευρώπη για τον τουρισμό και όχι άλλες υπήρους. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να καταστήσουμε περισσότερο γοητευτική, ας το πούμε στην Ευρώπη και θα πρέπει να σκεφτούμε τι γίνεται ακριβώς σαν ένα εσενιαίος χώρος πια η Ευρώπη για τουριστικό προορισμό ε, και έτσι να διευρύνουμε αυτή την αγορά για να μπορέσουμε όλοι μας να υποφεληθούμε. Ε, και πέρα από τον τουρισμό που παραδοσιακά ήταν ε, αντικείμενο ανταγωνισμού ανάμεσα σε περιφέρεια και περιφέρεια, στην ίδια χώρα και τα ίδια τα μέρη μια ενιαία περιφέρεια. Πρώτα απ' όλα λοιπόν που θα πρέπει να πετύχουμε είναι να τραβήξουμε νέου τουρίστε και μετά από τη στιγμή που οι τουρίστε αυτοί θα διαλέξουν την Ευρώπη θα υπάρχει δυνατότητα οι διάφορε χώρε κάθε χώρα ξεχωριστά να μπορέσει με τις σειρά να προσελκύσει τους τουρίστες αυτούς να πάνε και εκεί. Άρα λοιπόν όφελος οικονομικό και επίσης υποστήριξη στον ε, ανταγωνιστικότητα και διάφορα άλλα θέματα που προκύπτουν πολύ σημαντικά όπως την ποιότητα της ε, τουριστικής προσφοράς στην Ευρώπη να ξεπεράσουμε τώρα ιδέες που μας καταδικάζουν ουσιαστικά, δηλαδή αυτό τους, ε, μιας, της, του εποχιακού τουρισμού, μια ορισμένη περίοδο του χρόνου, λίγους μήνες το χρόνο. Αυτό σημαίνει για την απασχόληση, για την οικονομική ανάπτυξη αρνητικά φαινόμενα, αρνητικές επιπτώσεις. Άρα λοιπόν μακρύτερη τουριστική περίοδος, να το υποστηρίξουμε αυτό και έτσι και κοινωνικά, κοινωνικο-οικονομικά κλπ. Και σίγουρα εδώ αναφέρομαι στα γνωστά μας ε, να βοηθήσει η μεταφορά ε, κινητικότητα, γιατί εντάξει να φτάσουν οι τουρίστες, αν δεν μπορούν όμως να μετακινηθούν άμεσα και γρήγορα στην Ήπειρό μας, πώς θα μπορέσουμε να κερδίσουμε μπροστά σε αυτή την πρόκληση στην οποία αναφέρθηκα. Επίσης και η φορολογία είναι πολύ λεπτό το θέμα. Έχει να κάνει και με εθνικά συμφέροντα που είναι αντιφατικά και πολύ συχνά λέμε ότι θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε αυτά με ένα κλειδί ευρωπαϊκό και να αντιμετωπίσουν την πρόκληση. Και μέσα στην Ευρώπη θα πρέπει να υπάρχουν οι ίδιες αφετηρίες, ίδιες, τα ίδια που θα ισχύουν για όλους. Διαφορετικά διακινδυνεύουμε να χρησιμοποιήσουμε, να καταβάλουμε προσπάθειες ε, όπως πριν, ε, να κάνουμε κάτι το καινούριο και μετά να υπάρξει μια στρέβλωση του ανταγωνισμού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ορισμένοι θα υποφεληθούν και θα καταδικαστούν άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν απαιτείται η πτυχή αυτή να αντιμετωπιστεί κατάλληλα, αποτελεί ε, κάτι το σημαντικό και θα πρέπει να αποφύγουμε τις αντιπαραθέσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ορισμένα σημεία κλειδιά στα οποία μπορούν να βοηθήσουν και οι συνάδελφοι. Τώρα να δούμε τι εικόνα θα προσφέρει η Ευρώπη. Εμείς ε, σκεφτόμαστε μετά από πρόταση του Αντιπρόεδρου Ταγιάννη να έχουμε ένα, μια μάρκα, στην πούμε μια σφραγίδα Ευρώπη για να δείξουμε τι προσφέρουμε ακριβώς στις νέες αγορές που θα ανοίξουν και να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο και καλύτερα ένα σημαντικό εργαλείο, αυτό το Visit Europe κόμμα αυτό το, αυτή την ιστοσελίδα. Όχι, δεν το διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα ευρωπαϊκό όργανο, αλλά το ITC που είναι οι εθνικοί οργανισμοί τουρισμού των διαφορών χωρών. Και έχουμε και ένα πολύ σημαντικό θέμα ακριβώς πώς θα προσελκύσουμε ε, καλύτερα μέσω της κατάλληλης ε, βίζας, ε, εύκολης, γρήγορης και αυτό θα πρέπει να το δούμε και εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικότατο αυτό το θέμα και απέναντι σε χώρες όπως αυτές τις αναδυόμενες που είπα πριν έχουμε διαδικασίες που ισχύουν και διαφορετικό κόστος από τη μία χώρα στην άλλη για να εκδοθούν αυτές τις θεωρήσεις για την επίσκεψη των τουριστών τους. Θα πρέπει να θετήσουμε κοινέ διαδικασίες ώστε όποιο τουρίστας θέλει να έρθει στην Ευρώπη να είναι το πετύχει εύκολα και γρήγορα όπως και επίσης και οι tour operators. Ελπίζω να με βοηθήσετε και σχετικά με αυτά που είπα πριν και τις φραγίδες, τις ποιοτικέ φραγίδες, φραγίδα ποιότητας και αυτό που εμφανίστηκε και στη συζήτηση με τους και ηγητές είναι να αποφύγουμε ε, πολλά, πάρα πολλά σήματα που σαν τα μανιτάρια φυτρώνουν εδώ και εκεί και κάθε χώρα έχει τη δική του τη σφραγίδα και οι περιφέρειες μετά, πόλεις από εδώ από εκεί προωθούν ε, διάφορες δικές σφραγίδες ποιότητας και εντάξει περισσότερη προσφορά αλλά μειώνεται η αξία αυτής της σφραγίδας ποιότητας, αυτού του σήματος ποιότητας ε, και η εμπιστοσύνη επίσης ε, των ενδιαφερομένων. Λοιπόν, να υπάρχει κάτι κάτι, ένα ενιαίο σήμα, σαν ομπρέλα πάνω απ' ε, και ο καθένας να μπορεί να συμμετέχει εκεί, να το χρησιμοποιεί και έτσι μέσα σε μερικά χρόνια να έχουμε αυτό το σήμα ευρωπαϊκής ποιότητας που να δείχνει που υπάρχει αυτή η κατάλληλη τουριστική οργάνωση, να υπάρχει ένα κοινό επίπεδο ποιοτικό ε, και ο χρήστης να υποφελείται στο τέλος, ο τουρίστας δηλαδή και επίσης την ταξινόμηση των ταξιδοχείων, τα αστέρια. Αυτό συζητείται εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ε, από εδώ και από εκεί και στο κείμενο επανέλαβα ότι θα πρέπει να έχουμε τη διάθεση να προχωρήσουμε σε μια εναρμόνιση αυτού του συστήματος με τα αστέρια στα ξενοδοχεία και να επωφεληθούμε και από διάφορες θετικές εμπειρίες σε μερικά κράτη-μέλη ξεκινώντας από ορισμένα βήματα επαγγελματικών κλάδων που βοηθούν για κοινά πρότυπα για την ε, απονομή αυτών των αστεριών. Και επίσης ε, ο τουρίστας ακριβώς να ξέρει ακριβώς ε, πόσα αστέρια αντιστοιχούν σε ποια ποιότητα ε, και σε ορισμένες υπηρεσίες που να ισχύουν αυτά από τη Σικελία μέχρι τη Φινλανδία. Και ακόμα δύο σημαντικότατα θέματα εφαρμόζοντας ε, τη στρατηγική του 2020, την επαγγελματική κατάρτιση και τη νέα τεχνολογία. Χρειαζόμαστε να καταρτήσουμε κόσμο για τον τουρισμό που να μην είναι μόνο η κατάρτιση προσωπικού που έχει άμεση μόνο επαφή με τον ε, ε, τουρίστα δηλαδή, ο, το ξενοδοχειακό, το, το, το, υπάλληλο οι μπάρμαν και οι μάγειροι, θα πρέπει να είναι και οι υπόλοιποι που να τους καταρτίζουμε για να μπορέσουν να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα ροή των νέων αγορών στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως θα πρέπει ταυτόχρονα ιδιαίτερα να προσπαθήσουμε πάνω στο θέμα των νέων τεχνολογιών γιατί έχει αλλάξει ριζικά ο τρόπος ε, τουρισμού σχέση με το παρελθόν τώρα είναι μέσα και στο ίντερνετ. Ο κάθε τουρίστας πολύ συχνά μόνος του επιλέγει μέσω του ίντερνετ τι υπηρεσίες θέλει να έχει και για τη μεταφορά του, το ταξίδι του και τα πολιτιστικά, επιτόπου τα στοιχεία προσφέρουν και έτσι να υποστηρίξουμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας τις ευρωπαϊκές να δείξουν την ε, αξία τους τα όσα προσφέρουν εκεί στο ίντερνετ και είναι λοιπόν με ένα καινοτόμο τρόπο και όλα αυτά για να υποστηρίξουμε αυτή την ανταγωνιστικότητα των ε, ε, επιχειρήσεων μας τον τουριστικό και να έχουμε και μια πλατφόρμα νέα ευρωπαϊκή ICT και τουρισμού λοιπόν νομίζω ότι κάτι τέτοιο αποτελεί μια θετική πρωτοβουλία που θα πρέπει να υποστηρίξουμε για να εφαρμοστεί γιατί πάνω σε αυτό υπάρχει ένα κενό το αντιμετωπίζουν ε, ε, κάμποση ε, αλλά αρκετοί πάντως και ακόμη οι διάφορες μορφές τουρισμού και ολοκληρώνω εδώ. Ίσως το είδατε ήδη στο κείμενό σας ένα λεπτομερή κατάλογο. Θα ήθελα όμως να με βοηθήσετε με τις τροπολογίες σας να δώσω μια οριστική μορφή σε αυτό γιατί δεν μπορεί να μας δεν αρκέσει εντάξει ότι υπάρχει ε, ε, αγροτοτουρισμός ε, ε, γιατί του αρέσει η θάλασσα, που του αρέσει το βουνό κλπ. Αλλά θα πρέπει να υποφεληθούμε εδώ από την έκθεση αυτή, από την εργασία αυτή, πώς θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε διάφορες μορφές τουρισμού. Να δούμε και τους τομείς εκείνου που αναπτύσσονται ταχύτερα και περισσότερο. Τελευταίο, τελευταίο και μετά μπορούν να παρέμβουν οι συνάδελφοι, έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση. Το γνωρίζετε ασφαλώς οι δημοσιονομικές προοπτικέ και πάνω στον πολιτή προπολογισμό πάνω στον οποίο εργαζόμαστε τώρα ε, είχε ισχύσει αυτά όταν δεν υπήρχαν αρμοδιότητε για τον τουρισμό και τώρα οι πόροι είναι λίγοι, οι ειδικοί πόροι για τον τουρισμό και σε μεγάλο μέρος είναι κάπως ε, κρυμμένη αυτοί οι πόρη στο βάθος βάθος των διαρχοτικών ταμείων, το μείο συνοχής είτε το γεωργικής ανάπτυξης. Ε, θα πρέπει λοιπόν ε, ακόμα περισσότερο να φανούν αυτά, πιο διάφανα αυτά τα κονδύλια που μπορούν να πάνε, μπορούν να αποδοθούν εκεί και που βρίσκονται στα διαρχοτικά ταμεία και θα πρέπει να εργαστούμε και με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα ώστε ορισμένα σχέδια να υποστηριχθούν άμεσα με ειδικά προγράμματα λοιπόν λοιπόν και με ειδικά κονδύλια. Θα πρέπει να έχουμε την πιο φιλόδοξη δυνατή στρατηγική για τον τουρισμό, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι εκεί βέβαια και ορισμένα που δεν μας στοιχίζουν για την ανταλλαγή της βέλτιστης πρακτικής που εφαρμόζει ο καθένας, αλλά όμως άλλες πρωτοβουλίες απαιτούν κονδύλια, απαιτούν χρήματα και πολλές φορές πολλές ε, πολιτικές ομάδες ε, υποστήριξαν ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί έτσι ο τουρισμός γιατί θα πρέπει να δοθεί αυτή αυτή η μάχη στα πλαίσια της νέας δημοσιονομικής προοπτικής του 2014. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τώρα οι εκπρόσωποι των κομμάτων για την έκθεση και ξεκινάμε από τον κύριο Δανέλο που είναι των σοσιαλιστών παρακαλώ τουριστική βιομηχανία της Ευρώπης διέρχεται μια περίοδο καμπής. Για την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης και της ύφεση των οικονομιών των χωρών μελών μπορεί να συμβάλλει με την εξασφάλιση αλλά και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, διασφάλιση εσόδων στις τοπικές οικονομίες και ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη. Για να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας απαιτούνται μέτρα και πολιτικές συντονισμού, εναρμόνισης, επέκτασης, και ποιοτική αναβάθμιση του ευρωπαϊκού τουριστικού προϊόντος. Η πολυμορφία, η διαφορετικότητα, η πολυπολιτισμικότητα της Ευρώπης προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ανάπτυξη κάθε μορφής θεματικού τουρισμού. Η ανάπτυξη και προώθηση των μορφών του διαφοροποιημένου τουρισμού μπορεί να αποτελέσει τη μόνη αποτελεσματική απάντηση στις τρευλώσεις, τα προβλήματα και την υποβάθμιση που έχει οδηγήσει σε πολλές περιοχές το μοντέλο του ισοπεδωτικού μαζικού τουρισμού. Αυτό που έχει ανάγκη η τουριστική μας βιομηχανία είναι να περάσει από την εποχή της ανάπτυξης του τουρισμού στην εποχή του τουρισμού της ανάπτυξης. Η έκθεση του συναδέλφου Φιντάντσα εκφράζει σε πολύ μεγάλο βαθμό κοινέ προσεγγίσεις. Θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο στην πρώτη μας έκθεση ως Κοινοβούλιο για τον τουρισμό που αποτελεί πλέον ευρωπαϊκή πολιτική να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μερικές τουλάχιστον από τις 21 δράσεις που αναφέρονται στην ανακοίνωση ένα συγκεκριμένο σχέδιο εφαρμογής με ημερομηνίες και χρονοδιαγράμματα. Ένα σαφής προγραμματισμός θα επιτρέψει την ορθότερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών για την προώθηση των δράσεων που προτείνει η Επιτροπή καθώς επίσης και συγκεκριμενοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων και των πόρων που θα τις στηρίξουν. Προς την κατεύθυνση της ποιοτικής αναβάθμισης και της ανανέωσης του ευρωπαϊκού τουριστικού προϊόντος, πιστεύω θα βοηθούσε η εισαγωγή νέων αρχών, όπως οι αρχές της διαπεριφερειακότητας, interregionality, και της συμπληρωματικότητας, complementarity η αρχή της συμπληρωματικότητας συνεπάγεται τον αποκοινού σχεδιασμό με θεματικά και γεωγραφικά κριτήρια των εθνικών πολιτικών τουρισμού, παραδείγματο χάρη μοντέλων θεματικού τουρισμού ή συγκεκριμένων τομέων παροχής τουριστικών υπηρεσιών, ανεξάρτητα αν οι περιοχές αυτές συνορεύουν ή όχι. Η αρχή της διαπεριφερειακότητας συνδέεται με τον ενιαίο σχεδιασμό των τουριστικών υπηρεσιών είτε σε ενιαίο γεωγραφικά χώρο, παραδείγματος χάρη μεταξύ γειτονικών περιφερειών, αλλά και σε κοινή θεματική βάση μεταξύ διαφορετικών πιθανώς απομακρυσμένων περιφερειών. Στόχος της εισαγωγής των προτινόμενων αρχών στην υποδιαμόρφωση ευρωπαϊκή πολιτική τουρισμού είναι πρώτο η μεταφορά του πεδίου ανταγωνισμού που υπάρχει σήμερα μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής τουριστικής πολιτικής στο πεδίο του ανταγωνισμού μεταξύ της Ευρώπης και των τουριστικών προορισμών τρίτων χωρών. Δεύτερο, στη σημερινή συγκυρία της οξείας οικονομικής κρίσης ζητείται η δημιουργία αναπτυξιακού πλεονεκτήματος σε περιοχές τουριστικά υπανάπτυκτες σήμερα και φυσικά η περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού της Ένωσης με πιο ισόρροπη ωστόσο κατανομή του προϊόντος σε γεωγραφική και κοινωνικο-οικονομική κλίμακα προσφέροντας βιώσιμη περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά ανάπτυξη. Και τρίτο, φέρνουν τέλος επί της ουσίας κοντύτερα περιφερειακές αρχές και τοπικές κοινωνίες συμβάλλοντας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δούδης εκ μέρους των Φιλελευθέρων παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αποτελεί ιστορική ευκαιρία Ακριβώς επειδή μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας τώρα ξεκινάμε να μιλάμε για τον σαν αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν ξεκινάμε βέβαια από το μηδέν. Και ο προκάτοχός σας, ο κύριος Κώστα, κύριε Σίμψον, είχε επεξεργαστεί, είχε συντάξει ένα κείμενο που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή ιδιαίτερα δυνατή βάση για την σημερινή μας εργασία. Και μαζί με όλους τους εισηγητές με το Σταύρο και λοιπά και με άλλους συναδέλφους όλοι μας προσπαθούμε να δούμε, να πούμε ότι ο τουρισμός θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μοχλό ιδιαίτερο για την ανάκαμψη της οικονομίας της Ευρώπης στο σύνολό της. Ο τουρισμός δίνει το 5% του άμεσου ΑΕΠ, το 10% του συνολικού ΑΕΠ και έχουμε στον τομέα το 10% των πολιτών στην Ευρώπη που απασχολούνται στον τουρισμό αλλά για μας θα πρέπει να ανέβει ακόμα περισσότερο. Γιατί στην Ευρώπη έχουμε μία δυστυχώς ε, ε χειροτέρευση της καταστάσεως ε, στην Ευρώπη. Η γεωργία εγκαταλείπεται, ας πούμε, και ο τουρισμός θα μπορούσε να αποτελέσει τον πραγματικό μοχλό ανάπτυξης των επομένων δεκαετιών, των μελλοντικών δεκαετιών. Και είπαμε ότι για την Ευρώπη θα μπορούσε να είναι ο αιώνας του τουρισμού. Δεν το λέμε έτσι τυχαία αυτό, μόνο, για να το πούμε. Και απέναντι στρατηγική 2020 της Ευρώπης, ο τουρισμός έχει κάθε χαρακτηριστικό για να είναι το σύστημα που να δίδει αυτό που υιοθετήσαμε στην αρχή της ε, θητείας μας. Έχει και τα τρία βασικά χαρακτηριστικά. Είναι έξυπνος μοχλός ανάπτυξης, ε, είναι αηφόρος και επίσης συμπεριλαμβάνει πολλά και διάφορα στοιχεία. Είναι πλατής παράγοντας. Γιατί πλατής παράγοντας. Για πρώτη φορά τα 550 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών και γύρω στον κόσμο δεν έχουν πια σύνορα, δεν εμποδίζονται από κάτι. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε ιδιαίτερα, να συντάξουμε όσο γίνεται καλύτερα το κείμενό μας και εντάξει όλοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν δεν μπορεί να αποτελέσει το μοναδικό κείμενο στο οποίο θα αναφερθούμε στον, στον τουρισμό. Αποτελεί όμως ε, το πρώτο βασικό βήμα για να ανοίξουμε και άλλα περάσματα. Όπως είπε και ο Φιντάντσα πριν από λίγο, θα πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα να το αντιμετωπίσουμε το οικονομικό το πρόβλημα, αλλά επίσης και μια ολοκληρωμένη πολιτική τουριστική. Όταν μιλάμε για τον τουρισμό, μιλάμε για πολλούς και διάφορους τομείς που θα πρέπει να κινηθούν. Θα πρέπει να αποτελέσει σύστημα ο τουρισμός. Γύρω-γύρω από τον τουρισμό θα πρέπει να αναπτυχθούν όλοι οι υπόλοιποι τομείς, όπως η γεωργική παραγωγή, οι υπηρεσίες, οι μεταφορές να βελτιωθούν. Όλα αυτά από τη στιγμή που θα δώσουμε χώρο, θα κινηθούν όλα αυτά, θα δούμε ότι θα κινηθεί το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας και τα πολιτιστικά στοιχεία και γεωγραφικά τα διαμερίσματα όλοι μαζί θα ε, παρουσιάσουμε έτσι μια ενωμένη εικόνα της Υπήρους μας που είναι και ο κόσμος ολόκληρος, ε, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε για σκεφτείτε το η Κίνα θα ρίξει ένα εκατομμύριο πολίτες στην αγορά θα είμαστε έτοιμοι. Αυτό πρέπει να αποτελέσουν ε, ε, παράγοντα ανάπτυξης και όχι καταστροφής του περιβάλλοντος μας. Ε, θα πρέπει να αποτελούν λοιπόν βασικό στοιχείο σε αυτή την αηφόρα ανάπτυξη πάνω στην οποία εργαζόμαστε. Ένα πραγματικό εργαλείο για μια νέα Ευρώπη, για την οποία νέα Ευρώπη όλοι μας καταβάλουμε προσπάθειες. Ευχαριστώ κυρία Μπρέπερς εκ των Πρασίνων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φιντάντσα για την εξαιρετική του έκθεση. Σε αυτό το σχέδιο έκθεσης ξέρω ότι δούλεψε πάρα πολύ και είχαμε αρκετές επαφές στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της έκθεσης. Με ακούτε καλά? Μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα Ιταλικά, λέει ο Πρόεδρος εμφανίζεται ένα βουητό αλλά χωρίς καθόλου φωνή στην Ιταλική καμπίνα. Έχουν μόνο Ιταλοί πρόβλημα. Με ακούτε ακόμη. Δεν έχουμε διερμηνία στα Ιταλικά ή τώρα έχουμε. Νομίζω τώρα είμαστε εντάξει. Λοιπόν, έλεγα ότι ο κύριος Φιντάντσα έκανε αυτή τη θαυμάσια έκθεση. Θα τον ευχαριστήσω τώρα για τρίτη φορά λοιπόν. Ελπίζω να με ακούτε αυτή τη φορά. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. Σας ευχαριστώ και για τον ιδιαίτερα ανοιχτό τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την έκθεση αυτή και ε, τις επαφές που είχε με τους σκιώδεις εισηγητές. Όταν ξανακοίταξα την έκθεση την περασμένη εβδομάδα, αναρωτήθηκα μήπως θα ήταν προτιμότερο να έχουμε ένα πιο σύντομο κείμενο. Και το άκουσα και από άλλους συναδέλφους αυτό ως παρατήρηση. Μιλάμε για την μοναδική προστιθέμενη αξία που μπορεί να δώσει η Ευρώπη στον τουρισμό στο μέλλον με βάση το άρθρο 195. Εδώ στην έκθεση φαίνεται ότι συμπεριλαμβάνουμε όλα τα σημεία της ανακοίνωσης της Επιτροπής και δεν ξέρω μήπως ε, χάνουμε την ε, επικέντρωσή μας στους βασικούς μας στόχους. Γιατί το κείμενο μπορεί να γίνει ακόμη και περισσότερο μακροσκελές αν συμπεριλάβουμε και περισσότερες τροπολογίες. Στο παρελθόν το Κοινοβούλιο έχει ήδη ψηφίσει αρκετά ψηφίσματα για τον τουρισμό και θα πρέπει να αξιολογήσουμε και τα προηγούμενα ψηφίσματα, αντλώντας έμπνευση και από αυτά. Και αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τα πιο σημαντικά σχόλια που έχουμε εμείς από την ομάδα των Πρασίνων, που θα είναι και οι βασικές προτεραιότητες για τις τροπολογίες μας. Ο τουρισμό είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό οικονομικό τομέα, όπω είπαν πολλοί συνάδελφοι, αλλά θα ήθελα επίση να τονίσω πόσο μεγάλη ποιότητα προσδίδει ο τουρισμός στα θέματα εμπλουτισμού του πολιτισμού. Υπάρχει σαφώς μια κοινωνική διάσταση και ο τουρισμός μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο την οικονομία, αλλά και την γενικότερη ευημερία και πολιτιστική άνοδο. Όσον αφορά τα σήματα, είπε και ο εισηγητής ότι υπάρχουν πάρα πολλά σήματα και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να απλουστεύσουμε την κατάσταση σε σχέση με τα σήματα που θα υπάρχουν, γιατί δεν θέλουμε να προσθέσουμε νέα σήματα σε ένα μακρύ κατάλογο άλλων σημάτων. Πρέπει ένα καινούριο σήμα το οποίο θεσπίζουμε να είναι ξεκάθαρο και να έχει και νόημα. Επίσης πρέπει να προβλέψουμε και κάποιες κυρώσεις εάν τα προτινόμενα μέτρα δεν τηρούνται και να αναλύσουμε την προστιθέμενη αξία των σημάτων πριν δηλαδή δημιουργήσουμε νέα σήματα, να αξιολογήσουμε παλαιότερα σήματα και να δούμε τι θα προσθέσουν τα νέα μας σήματα. Να εξετάσουμε επίσης τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές, να προσπαθήσουμε να εναρμονίσουμε τις καλές πρακτικές όπου αυτό είναι δυνατόν και να λάβουμε υπόψη μας τα θέμα της αηφόρου ανάπτυξης και της προσβασιμότητας. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα σημεία και δεν μπορούμε να τα απομονώσουμε και να τα εφαρμόσουμε σε ορισμένους τομείς και μόνο. Θα πρέπει να διατρέχουν όλους τους τομείς και να αποτελούν εγγενές τμήμα μιας πολιτικής τουρισμού. Μιας πολιτικής που θα είναι βιώσιμη και στο μέλλον. Ο τουρισμός και βέβαια είναι συνδεδεμένος και με την κλιματική αλλαγή, διότι και προκαλεί επιπτώσεις στο κλίμα και υποφέρει από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Πρέπει λοιπόν να θεσπίσουμε εργαλεία τα οποία θα μας δώσουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε όλα τα σχετικά προβλήματα. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση τώρα και προς τον εισηγητή αλλά και προς την Επιτροπή. Δεν έχουμε νομοθετική εξουσία για να ζητήσουμε κάτι στον τομέα του τουρισμού. Ίσως όμως να υπάρχει δυνατότητα ενός χάρτη στον τομέα του τουρισμού που θα αποτελέσει μια καλή πρωτοβουλία. Ίσως κάτι τέτοιο να είναι εφικτό. Είναι μια ιδέα που την άκουσα από πολλούς και θα ήθελα να ακούσω και ποια είναι η γνώμη του εισηγητού και ποια είναι η γνώμη της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικό αυτό το σημείο. Ελπίζω να έχουμε το χρόνο να συντάξουμε τις τροπολογίες μας και να τις υποβάλουμε. Ευχαριστούμε κύριε Μπρόπελ. Σας άφησα ε, λίγο περισσότερο χρόνο γιατί ε, ξεκινήσατε με, μια τριπλή, με ένα τριπλό ξεκίνημα. Κυρία Φως τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, λέει η κυρία Φώστερ, να το ξαναδούμε λίγο κάνοντας ένα βήμα προς τα πίσω. Ξέρω ότι ο εισηγητής έχει καταβάλει μεγάλο κόπο, αλλά τη σταδιοδρομία μου σε μεγάλο βαθμό εγώ την έχω περάσει στον τομέα των μεταφορών και του τουρισμού και θα ήθελα να αντλήσω από την εμπειρία αυτή. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε και να μην παραβλέψουμε είναι ότι η αιτιολογική σκέψη Δέλτα είναι σαφής και λέει ότι θα πρέπει να συμπληρώνονται οι δράσεις ε, στα κράτη-μέλη από τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βλέποντας τις λεπτομέρειες της έκθεσης κάπως ανησυχώ γιατί είναι σαν να πρόκειται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευθύνει την πολιτική τουρισμού ή σαν να το, διευθύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή τέλος πάντων κάποιος ευρωπαϊκός φορέας μοιάζει να θέλουμε να διευθύνει τον τομέα του τουρισμού. Υπάρχουν βέβαια πολύ θετικά σημεία και πρέπει να ακολουθήσουμε μια θετική αντιμετώπιση βλέποντας ε, τι κάνουμε με τους κανονισμούς ε, για την υγεία και ασφάλεια παραδείγματος χάρη σε όλη την Ευρώπη, για την ίση μεταχείριση, για τα άτομα μειωμένης κινητικότητας, για την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων σε ολόκληρη την Ευρώπη για να διευκολύνουμε τη μετακίνηση, την ταχεία μετακίνηση των επιβατών και στι συνδρομικές μεταφορές όπως πολύ καλά γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε. Επίσης το θέμα της αμοιβαία αναγνώρισης προσόντων είναι και αυτό ένα σημαντικό ε, θέμα που έχει βοηθήσει ε, και όταν ε, βελτιώνουμε τέτοια στοιχεία βελτιώνουμε την κινητικότητα γενικότερα. Εδώ μιλάμε για εκατομμύρια πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη που κινούνται σε όλη την αλυσίδα των μεταφορών, των ξενοδοχείων, των υπηρεσιών. Επομένως έχουμε ένα αυξανόμενο οικονομικό τομέα και νομίζω ότι δεν υπάρχει στρέβλωση ανταγωνισμού. Όταν μιλάμε για τουρισμό, μιλάμε για ανταγωνισμό. Θέλουμε καλή ποιότητα, θέλουμε σωστές μεταφορές, επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται, ούτω ώστε ε, να μπορέσει να υποφεληθεί ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής θέλει ένα καλύτερο προϊόν. Μερικές φορές είναι δύσκολο να εναρμονίσουμε τα πάντα. Όταν θέλουμε να πάμε για σκι, μπορεί να μην θέλουμε να πάμε στην ε, Μάλαγκα. Χρειάζεται λοιπόν η δυνατότητα διαφοροποιημένου προϊόντος προς ε, τον πολίτη και κάθε χώρα μπορεί να προσφέρει κάτι διαφορετικό και αυτή είναι και η επιλογή η οποία προσφέρεται στους καταναλωτές. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει στρέβλωση ανταγωνισμού ακόμη να μην ξεχνάμε την επικουρικότητα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποφασίζουν. Να, μην, να προσέξουμε να μην καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου θα υπάρχουν υπερβολικές περιοριστικές ρυθμίσεις και υπερβολικές παρεμβάσεις. Δεν είναι δουλειά μας αυτή το να αρχίσουμε εμείς να επιβάλλουμε ρυθμίσεις στον τομέα του τουρισμού και όταν μιλάμε για ε, το ΦΠΑ, αυτά είναι εθνικές αποφάσεις, δεν έχουν καμία σχέση με τη δική μας Επιτροπή. Ακόμη θα πρέπει να προσέξουμε ε, κάποιες αναφορές που δεν είναι καθόλου αρμοδιότητα δική μας. Τα θέματα εναρμόνισης της πολιτικής θεωρήσεων διαβατηρίου και ομαδικές ε, θεωρήσεις διαβατηρίου δεν είναι καθόλου δική μας αρμοδιότητα αυτό το θέμα. Και υπάρχουν ε, και άλλα σημεία, η παράγραφος 12 και η παράγραφος 11. δεν είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνεργάζεται με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Μπορεί η Επιτροπή να έχει κάποια, κάποιες κατευθυντήριες γραμμές και κάποια πρότυπα, αλλά δεν είναι καθόλου δουλειά της Επιτροπής να συνεργάζεται με τους ε, ταξιδιωτικούς πράκτορες. Επίση σημείωσα αυτό που υπάρχει και ε, για την ε, ε, πύλη σε πολλές γλώσσες θα πρέπει να φροντίσουμε το κόστος να είναι λογικό, να μην αυξάνουμε το κόστος με τις δραστηριότητες που προτείνουμε. Σίγουρα υπάρχει πολύ σωστό περιεχόμενο στην έκθεση που μας προτείνει ο εισηγητής, αλλά νομίζω ότι ε, κάπως θα πρέπει να συγκρατηθούμε σε κάποιους τομείς για να δούμε κατά πόσο είναι πρακτικό και βιώσιμο και πώς να παραμείνουμε στην αιτιολογική σκέψη που διέπει το ρόλο μας με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας, ούτως ώστε να συμπληρώνουμε τις δράσεις κατών μελών και να μην ε, ε, προτρέχουμε και προκαταλαμβάνουμε αυτά τα οποία θα κάνουν τα κράτη-μέλη. Να μην ε, δηλαδή απομακρυνθούμε από αυτό το οποίο θέλουν οι καταναλωτές που είναι το να ταξιδέψουν και να μπορούν να δουν άλλες χώρες οι ταξιδιώτες θέλουν να βλέπουν διαφορετικά πράγματα και σαφώς εδώ το κόστος υπησέρχεται γιατί κάθε οικογένεια θέλει να μπορεί να συγκρίνει το κόστος ενός ταξιδιού στην Ευρώπη με το, τόξος, με το κόστος ενός ταξιδιού στη Φλόριντα. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι τον εισηγητή. Και πιστεύω ότι η συζήτηση αυτή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνάδελφοι, τρία λεπτά ο καθένα. ξεκινώ με την κυρία Ράνα, παρακαλώ, για τρία λεπτά μην υπερβάλλετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη όπως πάντοτε εξάλλου. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον κύριο Φιντάντσα για την έκθεσή του που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα γιατί και στην Επιτροπή Πολιτισμού έχουμε συνεργαστεί με τον συνάδελφο Φιντάντσα για το θέμα αυτό και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το θέμα του Ευρωπαϊκού Σήματος Ποιότητας και, το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. θέλουμε να έχουμε νέα στοιχεία όταν υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία προσφέρουν κάτι καινούριο για την Ευρώπη. Θα πρέπει να δούμε πού υπάρχουν κάποια ευρωπαϊκά σήματα ποιότητας και πού μπορούμε να προσθέσουμε κάτι παραπάνω με ένα σήμα ποιότητας το οποίο εμείς θα, θα προτείνουμε για να προσφέρουμε κάτι ενδιαφέρον προς τους τουρίστες ο στόχος της δουλειάς μας εδώ θα πρέπει να είναι το να δώσουμε κίνητρα στα κράτη-μέλη, να βελτιώσουν ακόμη καλύτερα τις τουριστικές τους υπηρεσίες και εκεί όπου δεν υπάρχουν τέτοιες υπηρεσίες να δημιουργηθούν τέτοιες τουριστικές υπηρεσίες. Υπάρχουν λοιπόν και γενικά σχόλια και πολύ συγκεκριμένα σχόλια όπως έκανε και ο συνάδελφος ο κύριος Φιντάντσα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ε, μια ισόρροπη στάση μεταξύ αυτών ε, των σημείων προς τα οποία μπορούμε να προχωρήσουμε και εκεί που δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και το πώς αυτό μπορεί να γίνει. Κάποιες παρατηρήσεις που έχω σημειώσει ως ε, λήψεις και τα οποία θα ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι ε, επειδή βρισκόμαστε σε περίοδο δημογραφικών ε, αλλαγών να φροντίσουμε ιδιαίτερα τα πιο ηλικιωμένα άτομα και να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία ε, στους τουρίστες Μεγαλύτερη ηλικία. και να δώσουμε τη δυνατότητα και στου ηλικιωμένους πολίτε να αποκτήσουν τη χαρά του ταξιδιού αν δεν γνωρίζουν αυτή τη χαρά ήδη. Ακόμη και το σύστημα εκπαίδευση και κατάρτιση είναι πολύ σημαντικό ούτω ώστε ε, ε, να αντιστοιχούν περισσότερο οι, υπηρεσίε. Σπουδέ ε, στον τομέα του τουρισμού, του τουρισμού με τι προσφερόμενε υπηρεσίε. Μας ενδιαφέρει βέβαια και η οδηγία για ε, τα οργανωμένα ταξιδιωτικά ε, πακέτα και ε, έχει ήδη ανακοινώσει η Επιτροπή το σχέδιο οδηγίας ε, εδώ και πολύ καιρό και θα ήθελα να ζητήσω να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν σε αυτήν την οδηγία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Δεγκράντες. Τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Φιντάντσα, σας ευχαριστούμε και το λέω επισήμω αυτό. Είναι υπέροχο αυτό. Και από τα σημεία κλειδιά είναι το είστε Ιταλό. Και έχετε ιδιαίτερη αρμοδιότητα. Αλλά η πύρα είναι ο ίδιος, η ίδια πύρα αποτελεί βαθμό και ένας Ιταλός είναι ο αρμόδιος και στην Ισπανία ας πούμε είναι πρώτη βιομηχανία της χώρας. Άρα λοιπόν ξέρουμε γιατί μιλάμε και δεν είναι εύκολη έκθεση. Αυτή η νέα αρμοδιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο τουρισμός μέσω της 195 ε, άρθρου της ε, Συνθήκης της Αβώνας, απαγορεύει την αρμόνιση και ίσως θα πρέπει να κολλιάνουμε τις γωνίες όπως είπε και ο συνάδελφος δεν θα πρέπει να μπούμε σε ξένα χωράφια εδώ πρόκειται για μια σοφή θέση αυτή της Λισαβόνας. Είναι πηγή πλουτίου για τις χώρες και διαφοροποίηση είναι κάτι το ελκυστικό. Και αυτή η αρμοδιότητα είναι ο κινητήρας της επιτυχίας. Περισσότερο ελκυστική στο σύνολό της Ευρώπη, χωρίς να βλάψει την εργασία των αγορών, των ε, χωρών ε, τις πρωτοβουλίες τους για να παρουσιάσουν τη, διατηχώρη τη τους. Ο καθένας ε, έχει δίπλα του, όχι μόνο φίλο όμως σαν χώρα, αλλά και ένα ανταγωνιστή. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα πετύχουμε αυτή την προστιθέμενη αξία. Και εδώ όλα όμως αυτά αναφέρονται δεν έξυπνα, ότι έχει σημασία το σήμα Ευρώπη ποιοτική. Θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα να μην διακινδυνεύσουν και άλλες αποδειγμένες αξίες και θα πρέπει να προσθέσουμε νέες δυνατότητες και όχι να βλάψουμε τις παλιές. Εδώ λοιπόν ε, νομίζουμε ότι σέβεστε αυτό το διαφορετικό χαρακτήρα του κάθε κράτους και με τη δυνατότητα ενός σχεδίου για καλύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση σαν πρώτο στόχο προορισμό τουριστών στον κόσμο και στις προτάσεις ε, είναι, οι προτάσεις του εισηγητού μας βρίσκουν σύμφωνος. Βέβαια θα διατυπώσουμε διάφορες συμπληρωματικές ε, των θέσεών σας προτάσεις και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την απεθνικοποίηση. Θα πρέπει να αποφύγουμε τις αντιθέσεις και επίσης ε, την ε, χαμηλή περίοδο και την υψηλή περίοδο για τον τουρισμό που βλάπτει τον τουρισμό. Να δούμε τον κοινωνικό τουρισμό. Έχουμε ιδιαίτερη σημασία που αποδίδουμε στην Ισπανία σε αυτό και να μπορέσουμε όλα αυτά να τα εφαρμόσουμε και με τον τουρισμό τρίτη ηλικία, ας πούμε και για ε, μεθοριακά και στην ίδια τη χώρα μας. Εδώ έχει σημασία η τρίτη ηλικία κύριε Πρόεδρε και ολοκληρώνω στην Ισπανία είναι οι Γερμανοί και οι Βρετανοί συνταξιούχοι καλύτεροι πελάτες μας και είναι ο καλύτερος κοινωνικός τρόπος έτσι να τους ευνοήσουμε που δεν έχουν τόσες δυνατότητες να μπορέσουν να μετακινηθούν ε, με τα μέσα που διαθέτουν μέσω της σύνταξή τους και ταυτόχρονα έτσι βοηθάμε και τις θέσεις τουρισμού στη κάθε χώρα και θα συντάξουμε ε, Ακριβώ τροπολογίε, αλλά ήδη η έκθεση νομίζουμε ότι είναι συνταγμένη με καλό και άριστο τρόπο. Ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, κάθε συμφωνία έχει μερικά θετικά στοιχεία. Και αυτό ισχύει και για τη συνθήκη τη Λισαβόνα βεβαίω. Όταν φτάσουμε στον τουρισμό όμω, ξέρετε, η Λισαβόνα, γύρω δεν θα εξυπηρετηθούμε κάλλιστα. Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι στο εθνικό επίπεδο ο τουρισμός είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Μπορείτε κάλλιστα να έχετε ένα πολύ καλό μπραντ για τη Σαρδινία, δηλαδή ένα καλή μάρκα και επίσης για την Ολλανδία κλπ. Πολύ ωραία αυτά. Άρα τι γίνεται με αυτό εδώ τη μάρκα θα λέγαμε των εισαγωγικών τι γίνεται με τον πολιτισμικό τουρισμό. Δεν πιστεύω πραγματικά πού βρίσκεται αυτή η αλήθεια, πού βρίσκεται αυτή η κατάσταση, διότι βλέπετε για κάθε παράγραφο θα πούνε χιλιάδες τροπολογίες καθότι αυτή τη στιγμή δεν είναι της Ευρωπαϊκής Αρμοδιότητας αυτό το θέμα και θα ψηφίσω κατά διότι δεν έχει σχέση με ό,τι προσπάθεια έχει κάνει ο κ. Φιντάντσο εισηγητής μου για αυτό το θέμα. Ο κύριος Μπάτσι είναι ο επόμενος παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον συνάδελφο Φιντάντσα για την εκθεσή του. Χρησιμοποίησε την ευκαιρία που μας δίδεται μέσω αυτού του νέου πολιτικού πλαισίου και των αρμοδιοτήτων αυτών. Χρησιμοποίησε λοιπόν την ευκαιρία για να μας ετοιμάσει αυτήν την πολύ καλή έκθεση. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον αυτές τις προειδοποιήσεις πολλών συναδέλφων ότι ε, εισάγουμε πάρα πολλές ε, περιοριστικές ρυθμίσεις. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα εάν προσπαθούμε να έχουμε κάποια εναρμόνιση σε κάποιους τομείς, όπως να έχουμε ταξινόμηση τη εκπαίδευση και κατάρτισης, παραδείγματο χάρη. Αυτό θα δώσει προστιθέμενη αξία στην Ευρώπη στον τομέα του τουρισμού. Ακόμη θα βελτιώσει και το νομικό πλαίσιο, όπως είπε ο κ. Φιντάντσε και αναφέρθηκε και η κυρία Ράνερ σε αυτό ε, και στην οδηγία για τα τουριστικά πακέτα, παραδείγματο χάρη γιατί συχνά ακούμε το θέμα των τουριστικών πακέτων και πιστεύω ότι θα ήταν καλή ευκαιρία που θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε κάποιες ε, ρυθμίσεις. Όσον αφορά τη δημογραφική ανάπτυξη, πιστεύω ότι θα, δίνουμε όλο και μεγαλύτερη σημασία στην υγεία. Επομένως, ο ιαματικός τουρισμός ε, είναι ένας τομέας που πρέπει να προσέξουμε. Εδώ θα έπρεπε να υπάρξει κάποιο είδους εναρμόνιση, γιατί υπάρχουν πολλές φορές αμφίβολες, ε, οι αμφίβολες ποιότητας υπηρεσίας. Και στο σημείο 11, εκεί που αναφέρονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό που αναφέρεται για την αλυσίδα ψηφιακής προσφοράς. Αν μπορεί ο συνάδελφος Φιντάντσα να μου το εξηγήσει. Και για τη δραστηριότητα των εθελοντών επίσης θα ήθελα να πω ότι και στον τομέα του τουρισμού σίγουρα θα είναι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη η δραστηριότητα των ε, εθελοντών Χρειάζονται όμως πολλές γνώσεις για την εξυγίανση και για τη βελτίωση ε, κάποιων τουριστικών περιοχών. Επομένως δεν αρκεί η δραστηριότητα των εθελοντών για κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κουμουτσάκος. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, η τουριστική βιομηχανία ήταν ε, πάντα μια πολύ σημαντική οικονομική δράση. Στην παρούσα εξαιρετικά δυσχερή οικονομική περίοδο αποκτά ακόμα περισσότερη βαρύτητα και σημασία. Γι' αυτό θα έλεγα επιτέλους έχουμε συγκεκριμένη θεσμική βάση για να μιλήσουμε και να δουλέψουμε για την ευρωπαϊκή πολιτική τουρισμού. Συγχαίρω τον συνάδελφο κύριο Φιντάντσα για το σχέδιο που μας παρουσίασε. Δεν θα είχα καμία δυσκολία να προσυπογράψω το σύνολο των όσων αναφέρονται σε αυτό το κείμενο. Θα ήθελα μόνο να, να αναφερθώ επιγραμματικά στα ιδιαίτερα θετικά σημεία του. Και λέω ναι στην τεχνολογία ναι, ναι στην ανάγκη δημιουργίας μιας πλατφόρμας για την τεχνολογία της πληροφορήσης και του τουρισμού, είναι παράγραφος 11. Λέω ναι στο Ευρωπαϊκό Σήμα για τον Τουρισμό Ποιότητας, είναι η παράγραφος 15. Λέω επίσης ναι στην ενίσχυση του αγροτοτουρισμού, γιατί βελτιώνει την ποιότητα της ζωής και τις ευκαιρίες για την οικονομία της υπαίθρου, είναι η παράγραφος 30. Λέω ναι στη δημιουργία ειδικού προγράμματο για τον τουρισμό στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών 2014-2020, η παράγραφος Τέλο, λέω ναι στη δημιουργία ειδική τεχνική ομάδα για τον τουρισμό στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, κλείνω με δύο γενικέ παρατηρήσει. Θα πρέπει πράγματι, και ακούστηκε από άλλου συναδέλφου, να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο θέμα τη επικουρικότητα. Η ευρωπαϊκή πολιτική τουρισμού θα πρέπει να επηρεάσει προ θετική κατεύθυνση τι εθνικέ πολιτικέ τουρισμού και όχι βέβαια να τι υποκαταστήσει. Και δεύτερη και τελική παρατήρηση πιστεύω και εγώ όπως ακούστηκε προηγουμένως ότι θα πρέπει να πιέσουμε την επιτροπή ώστε να προσδιορίσει το συντομότερο δυνατόν ένα χρονοδιάγραμμα, ένα road map καθώς και το περιεχόμενο για τις 21 δράσεις που έχει προτείνει για τον τουρισμό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χέγγεντς. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρόεδρε και χαίρομαι πραγματική ότι δώσατε αυτό το νόημα το οποίο είπατε προηγουμένω για μένα. Έτσι όπως το εκλάβατε. Καταρχήν θα ήθελα να πω το εξή. Λέγεται αυτή η επιτροπή τουρισμός και μεταφορών. Αλλά με τον τουρισμό δεν ασχολούμαστε. Μόνο με τις μεταφορές ασχολούμαστε. Νομίζω πραγματικά θα πρέπει να είναι περιφερειακή ανάπτυξη μέσα. Νομίζω πως λοιπόν ότι υπάρχουν βασικά σημεία τα οποία για να δούμε πραγματικά πώς θα πρέπει να το δούμε αυτό το δρόμο, ότι θα είναι βιωσιμότητα, να υπάρχει φορολόγηση, να υπάρχει ανταγωνιστικότητα, εναρμόνιση κλπ. κλπ τα οποία θα πρέπει. Συμφωνίζω λοιπόν με τον εισηγητή για όλα αυτά τα οποία είχε πάει, ιδιαίτερα σαν αυτό τον προπολογισμό και βεβαίω είναι το τελευταίο σημείο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στα διαστατικά ταμεία και στον προπολογισμό για αυτή. Και δεν νομίζω ότι πραγματικά αναφέρεται πολύ στον τουρισμό. Νομίζω πω πραγματικά είναι ένα πολύ καλό έργο ε, εργασία. Αυτό το οποίο μα χρειαζόμαστε δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή. Είναι έγγραφο. Είναι να γίνει το πράγμα. Στα, είναι τις αρμοδιότητες των κρατών μελών αυτών. Σαν ΕΕ λοιπόν, είμαστε, εμείς είμαστε πάρα πολύ ελκυστικοί. 27 χώρες αυτή τη στιγμή, 27 γλώσσες, διαφορετικές κουλτούρες. Είναι μοσαϊκό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτή είναι η δομή που υπάρχει. Δεν είμαστε τι έχουμε μετά από εκεί, Νέο Ζηλανδία, Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική κλπ. Ινδία, Κίνα κλπ. Νομίζω ότι το μοσαϊκό είναι αυτή τη στιγμή μόνη η Ευρώπη. Σε αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε ιδιαίτερα. Και ένα πράγμα το οποίο ελέγχθηκε επί δεν είναι αυτή τη στιγμή να καραμίζουμε τα πράγματα κάνοντας διάφορους κανονισμούς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο λοιπόν είναι καλό ξεκίνημα και νομίζω πραγματικά έκανε μια εξαιρετική εργασία. Είναι ασχέδιο βεβαίως εφόσον πραγματικά υπάρχουν τροπολογίες νομίζω πως πραγματικά τα πράγματα. 17 Μαρτίου στην Fifth Avenue έχει, θα κλείσει όποιος, θα κλείσει όλες οι υπότες γιατί είναι η μέρα του Σεν Πάτρικ Υπάρχει 40 εκατομμύρια το οποίο είναι Ιρλανδοί στην Ελλάδα. Και αυτό δείχνει πραγματικά πόσο κοσμο υπάρχει αυτή τη στιγμή και νομίζω πως πραγματικά μπορούμε σε αυτό το πράγμα να του ευχήσουμε. Είμαστε αυτή, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή σε ποια κατάσταση βρίσκονται η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ελλάδα κλπ. Ένα λοιπόν από τα στιγμή του οικονομική οικονομία είναι η, και ο τουρισμό πραγματικά, αλλά δυστυχώ αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αξιοποιήσει τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα έβαζαν σε αξία, θα αξιοποιήσουν αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ λοιπόν κύριε Φινάντσα για την προσπάθεια που κάθε και το σχέδιο το οποίο μα υποβάλλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Αστάρα παρακαλώ. Κυ... Κυρία παρακαλώ. Σα ευχαριστώ κάθε ευχή και συγχαρτήρια στον εισηγητή ιδιαίτερα πλήρης έκθεσης και με καλή αντιμετώπιση στον τουρισμό των σημείων κλειδιών. Οι άξονες ακριβώς είναι πάνω στην αρμοδιότητα, την αγωνιστικότητα, στην καινοτομία, πέρα από από υψηλές και χαμηλές τουριστικές σεζόν εποχές και επίσης ε, την κατάλληλη μετακίνηση. Ε, μεταφορές αυτές παίζουν ιδιαίτερη σημασία. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε τουρισμό, αν, ε, κυρίως αν μιλάμε για τα νησιά, τα περισσότερα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και τα βουνά βέβαια. Ε, στα νησιά υπάρχει πολλής τουρισμός, βασίζονται στον τουρισμό και ε, εγώ έρχομαι από τις Βαλεαρίδες νήσους και οι Βαλεωρίδες ε, είναι ε, καλύτερο συνδεδεμένο μέρος με τη Γερμανία και χάρη σε αυτές τις συνδέσεις ε, μπορούμε να μεταφέρουμε σε ένα εκατομμύριο κατοίκους δύο εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μια τροπολογία ίσως για να ενισχύσουμε τη βελτίωση αυτών των συνδέσεων με τις ορεινές και τις νησιωτικές περιοχές και να μπορέσει έτσι να ε, ενιοποιηθεί αυτός ο χώρος. Άλλωστε αναφέρεται και, ο, και η συνθήκη της Αβώνας. Επίσης μια αναφορά στις ε, παράκτιο τουρισμό και στις αγροτικές, επαναλαμβάνω, και ορεινές περιοχές. Και για το θέμα των σημάτων, εντάξει, θετικό, αλλά να είναι κάτι συμπληρωματικό των εθνικών πολιτικών και να υπάρχει ένα ειδικό σήμα του καθενός και να μην ε, επαναλαμβανόμαστε ας πούμε για την ποιότητα και άλλα υπάρχει και τη UNESCO το σήμα που πολλές περιοχές είναι γνωστές με αυτό το σήμα της UNESCO αλλά λοιπόν να μην το επαναλάβουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πούμε ότι αυτά είναι πολύ σημαντικά πολύ ενδιαφέροντα ίσως θα πρέπει όμως να κάνουμε κάτι ε, για να μπορέσει να συμμετάσχει κατάλληλα και ο κλάδος ε, θα πρέπει να βοηθήσει και για τις ε, μακρύτερες περιόδους ε, στις Βαλεαρίδες ε, έχουμε τα 2 εκατομμύρια τουρίστες μέσα σε τέσσερις μήνες. Καταλαβαίνετε την πίεση. Γι' αυτό θα πρέπει να επιμηκηθεί ακριβώς αυτή η περίοδος. Και καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται και άλλες μορφής ε, τουρισμός, εναλλακτικό τουρισμός ε, και ε, ας πούμε με τους συνταξιούχους που διαθέτουν χρόνο, έχουν χρήματα τη σύνταξή τους, γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα. Και ακόμα για τα άτομα με ε, διάφορα κινητικά και άλλα προβλήματα. Η Γερμανία είναι η πρώτη σε αυτά που βοηθάει και θα πρέπει λοιπόν να μπει και για τα άτομα με ειδικά προβλήματα, πώς θα βοηθούν για τον τουρισμό. Γι' αυτό λοιπόν, εναλλακτικό τουρισμό. Επίση, ο ναυτικό τουρισμό, σημαντικό τουρισμό ε, υψηλή ποιότητα, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται να δούμε και διάφορες περιπτώσεις ε, γιατί για να νιολογηθεί ένα σκάφος αυτό δημιουργεί προβλήματα. Θα πρέπει να δούμε πώς θα επωφεληθούμε αντίθετα. Εντάξει και πάλι συγχαρτήρια στον εισηγητή και θα συμμετάσχουμε με τροπολογίες για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και να τονίσουμε διάφορες πτυχές του κειμένου. Πάντως σίγουρα πρόκειται για ένα αξιόλογο κείμενο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τέιλερ έχει παρακαλώ το λόγο. Βρήκα το κουμπί. Ευχαριστώ. Την τελευταία εβδομάδα είχα μιλήσει επισκεπτόμενος την Δυτική Αγγλία και από τις αρχές εκεί τις τοπικές, τα εθνικούς, εθνικούς δρυμούς, σε εθνικού δημού, καθώς επίσης τους πράκτορες εκεί. Ξέρετε, πήγαμε στα Bed Breakfast και είδαμε πολλά πράγματα και τρία πράγματα ήρθαν στο μυαλό μου. Το πρώτο πράγμα το οποίο παρακολουθούσα είναι η σημασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή των μεταφορών για να υπάρξει ένας βιώσιμος τουρισμός. Και έχουμε ένα κεφάλαιο αυτή τη στιγμή για ένα βιώσιμο τουρισμό. Πρέπει να είμαστε πραγματικά μεγάλες προσπάθειες να μην αγνοήσουμε βεβαίως και να ψάξουμε να βρούμε την προστασία το, της επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος εκεί που θέλει να πάει ο κόσμος και να τον επισκεφτεί καθότι θέλει να πάνε εκεί να επισκεφθούν γιατί υπάρχουν ιδιαίτερες ομορφές, ιδιαίτερες ποιότητες και δεν θα πρέπει αυτή τη στιγμή να το υποσκάψουμε αυτό με μεγάλο τράφικ το οποίο θα δημιουργηθεί εκεί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι το πρόγραμμα λιτότητά, το οποίο ξέρω πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή πολλές υπάρχουν χώρες που κάνουν αυτό, αλλά και στην Ηνωμένο Βασίλειο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, και υπάρχουν περικοπές, περικοπές για τη δασοκομεία, η οποία ασχολείται με τα φορεία και αυτό περικόπει κατά 25%. Ο τουρισμός λοιπόν στη νοτιοανατολικά επίσης κόπηκε κατά 25%. Οι τοπικές αρχές λοιπόν αυτή τη στιγμή βλέπουν ότι υπάρχουν στο Isle of Wild, στο νησί του Wild αυτή τη στιγμή. Ε, ο κόσμος θέλει πάρα πολύ να πάει εκεί για τουρισμό, αλλά έκλεισαν τα πάντα και οποιαδήποτε πληροφορία το υπάρχει αυτό το νησί. Το, δεύτερο ακόμη πράγμα, το τρίτο μάλλον θέλω να πει, είναι ότι να υπάρχει αυτή τη στιγμή βοήθεια η οποία θα πράγματα με κατάρτιση, και οι οποίοι περιγράφονται εδώ στο σημείο 25. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει αυτό να συμβεί, διότι θα πρέπει όχι να αντικαταστήσουμε αυτή τη στιγμή τις επιδοτήσεις που είναι το κράτος, αλλά θα πρέπει όλοι αυτοί που εργάζονται εκεί να μπορέσουν να έρθουν. Νομίζω πως πραγματικά αυτά είναι τα τρία σημεία τα οποία ήθελα να σας υποβάλω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίσκεψή μου. Ευχαριστώ. Πριν εδώ στο Κομισιό. Καταρχήν εγώ θα ήθελα να πω στον ε, εισηγητή ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσπάθεια την ΟΠΑΝΕΛ και την καταπληκτική έκθεση που μας υποβάλλατε. Νομίζω πως είναι ενδελεχής η έκθεσή σας και νομίζω πως πραγματικά περιλαμβάνει πολλές εργασίες όπως έχουν γίνει μέχρι τώρα και πιστεύω ότι Υπάρχουν περικοπέ οι οποίε έχουν γίνει από το Κοινοβούλιο βεβαίω και για αυτέ. Αλλά αυτό που είπε ο κύριο Χέγγεν, και θα το επαναλάβω και εγώ, είναι πολύ σωστό. Καλούμεθα αυτή τη στιγμή μεταφορών και τουρισμού και ασχολούμε, δεν ασχολούμεθα πολύ με τον τουρισμό και δεν δίνουμε το χαρακτήρα στον τουρισμό που πρέπει, μια προτεραιότητα δηλαδή που θα πρέπει να έχει και τι χρειάζεται να υπάρχει αυτή, γιατί δεν υπήρχαν μέχρι τούδα αρμοδιότητες μας δίδονται. Ακόμη και αυτή τη στιγμή έχουμε περιορισμένες αρμοδιότητες για αυτό το θέμα. Λόγω της συμφωνίας και συμφωνώ με αυτό που ολέχθη προηγουμένως για τη συνθήκη όσον αφορά τη συνθήκη. Βεβαίω μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Πιστεύω όμως είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να, να δώσουμε πραγματικά μια όθηση στον τουρισμό καθότι όπως είπαν όλοι και ο κ. Δεγκράντας και άλλοι και το υπογράμμισαν νομίζω ότι για πολλέ χώρε αυτή είναι μια βιχανία πάρα πολύ σημαντική αποτελούν την ραχοκοκαλιά θα λέγαμε ορισμένων χωρών και χρειαζόμαστε να δούμε κύριε Φινάντζα, τι, να δούμε ποια, τι ακριβώς κάνει η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς για αυτό το θέμα διότι θέλω πάρα πολύ αυτή τη στιγμή να πληροφορηθώ για αυτό το θέμα και θα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι θα γίνει μια αναθεώρηση αυτής της οδηγίας που υπάρχει ως αυτόν τον, τουρισμό. Προηγουμένως δεν το είχε ακούσει κανένας αυτή τη στιγμή, αλλά ξέρετε ήταν το EasyJet και άλλα τα οποία ε, μεταφέρουν. Ε. Νομίζω πως αυτή είναι η θεώρηση η οποία θα γίνει. Θα πρέπει εμείς να, είμαστε, να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία η οποία γίνεται. Και τέλος, αυτό που θέλω να πω, έχετε δίκιο διότι πέρασε πάρα πολύ καιρό αυτή τη στιγμή όσον αφορά τη βιώσιμη μεταφορά όσον αφορά τον τουρισμό και βεβαίως υπάρχουν λόγοι οι οποίοι άπτονται τις ιστορίες, τις θρησκείες κλπ, κλπ, κλπ. Αλλά θα πρέπει να δούμε περισσότερο το ιστορική πλευρά και την ιστορική παράδοση αυτή τη στιγμή η οποία υπάρχει. Και είναι ένα σημείο το οποίο άρεσε πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα λόγο, αλλά επίση πάρα πολύ βοηθάει σε αυτέ τι περιοχέ, οι οποίε είναι με βιομηχανική περίοδο που έχει παρακμάσει η βιομηχανία για να ανακάμψουν από την οικονομική κρίση την οποία ε, υφίστανται. Ευχαριστώ πάρα πολύ και βεβαίω θα υπάρξουν τροπολογίε για αυτά. Ο κ. Όρτουν, κ. Επιτροπής, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά την ανταλλαγή σχολείων από πολλού ε, ευρωβουλευτέ, θα ήθελα εγώ απλώ να παρεμβώ για να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, καλή έκθεση την οποία μας παρουσίασε σήμερα. Και ε, απλώς θέλω να πω ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως φαντάζεστε, ε, τώρα μόλις αρχίζουμε την επεξεργασία αυτών των αξώνων που υπάρχουν στην ανακοίνωση. Και αυτό τηρώντας βεβαίως πλήρως αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στη συνθήκη της Λισαβόνας. Υποστηρίζουμε τη συμπληρωματικότητα και το συντονισμό στο επίπεδο που μπορούμε εμείς να δράσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν προωθούμε εναρμόνιση εθνικών ε, νομοθεσιών. Αυτό είναι ξεκάθαρο στη συνθήκη και δεν θα υποβάλουμε κάποια πρόταση προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης, ε, είμαστε ε, πρόθυμοι να επικεντρώσουμε τους πόρους μας στις πρωτοβουλίες εκείνες που έχουν προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή τουλάχιστον σε επίπεδο περισσότερων κρατών μελών. Προωθούμε λοιπόν αρκετές τέτοιες ε, πρωτοβουλίες και δεν θέλω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Υπάρχει η πλατφόρμα της ε, τεχνολογίας ε, πληροφορικής και επικοινωνιών, επίσης για τις τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μια προσπάθεια αποτύπωσης των δεξιοτήτων και προσόντων. Ε, ε, θα συνεργαστούμε με το Συμβούλιο της Ευρώπης και την UNESCO στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς για να μπορέσουμε να προάγουμε την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς ε, να υπάρχει επικάλυψη με τα σήματα που ήδη υπάρχουν στο επίπεδο της UNESCO. Επίσης, συνεργαζόμαστε με όλους τους εμπλεκομένους, προσπαθώντας να εντοπίσουμε μία προσέγγιση από τη βάση προς τα πάνω σχετικά με την προστιθέμενη αξία που θα μπορούσε να δώσει ένα ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας και θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε πώς αυτό το ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας μπορεί να υποστηρίξει και να συμπληρώσει τα σήματα που ήδη υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Θα έχουμε κάποια κοινά κριτήρια και μάλιστα θα γίνει ένα workshop στις Βρυξέλλες, ένα συνέδριο δύο ημερών όπως γνωρίζει ο κύριος Φιντάντσα. Συνεργαζόμαστε επίσης ε, με την ETC, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών και με τους Εθνικούς Οργανισμούς ε, Τουρισμού για να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε την Ευρώπη ως ε, ένα σύνολο προορισμών με μεγάλη πολυμορφία και προσπαθούμε να επικαιροποιήσουμε την υφιστάμενη πύλη Visit Europe και επίσης ε, κάτι που έχουμε ήδη ξεκινήσει να κάνουμε είναι ότι ε, αναπτύσσουμε και εδώ αναφέρομαι σε μια πρόταση της κυρίας Μπρέπελς ε, για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για υπεύθυνε επιχειρήσεις τουρισμού και υπεύθυνου τουρίστες. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό το θέμα, προσπαθούμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό χάρτη προς αυτή την κατεύθυνση βασιζόμενοι πάνω στη διεθνή ιδεοντολογία που υπάρχει για αυτό το θέμα. Θέλουμε να έχουμε ε, κάτι παραπάνω σε σχέση με τον βιώσιμο τουρισμό που έχουμε εδώ και ε, τρία χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με υποστήριξη του Κοινοβουλίου και να προωθήσουμε αυτές τις δραστηριότητες σε πιο τομεακό επίπεδο επικαιροποιούμε και το σχέδιο υλοποίησης που συζητήθηκε στη Μάλτα στο Φόρουμ των ευρίού και εδώ έχουν συνεισφέρει και τα κράτη-μέλη και πολλοί ιδιώτες φορείς, ε, ε, ιδιωτικοί φορείς και θα έχουμε μια επικαιροποιημένη ε, μορφή πριν από το Πάσχα όλα αυτά λαμβάνοντας υπόψη και ε, αυτά τα οποία έχουν να συνεισφέρουν ε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι και σε εθνικό και σε ιδιωτικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο. Προσπαθούμε να προωθήσουμε τον βιώσιμο και αηφόρο τουρισμό, λαμβάνοντας υπόψη, όπως σας είπα, την κοινωνία των πολιτών, ε, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους κοινωνικούς εταίρους, όλους τους πυλώνες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ε, τον τουρισμό κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πυλώνα τους λαμβάνουμε υπόψη ε, συμπεριλαμβάνοντας και την πολιτιστική παράμετρο και ε, τη δεοντολογία. Παραμένουμε σε στενή συνεργασία με όλους τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και από ό,τι άκουσα από τη συζητήσεις σήμερα αλλά και από την έκθεση είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε και την υποστήριξη του Κοινοβουλίου προς την κατεύθυνση προς την οποία κινούμεθα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Όρτον. Κάρλο θέλεις να προσθέσεις κάτι. Ε, ναι πρόεδρε ευχαριστώ και σύντομα. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, για την υποστήριξή τους, για τη βοήθεια τους στην τόσο σημαντική που μου πρόσφεραν. Να πω μερικά πράγματα στα γρήγορα. Το πρώτο αυτό το φάντασμα που περιπλανιόταν στις παρεμβάσεις πολλών συναδέλφων που μου θυμίζει την παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας. Μήπως υπήρξε κάποιο πρόβλημα με την διερμηνία και δεν με καταλάβατε κανένα από τα άρθρα που έγραψα εγώ, που σύνταξα εγώ, δεν έχει, δεν περιλαμβάνει κάτι που να παραβιάζει αυτή την αρχή της επικουρικότητας. Εγώ ήθελα να εντάξω το κείμενο αυτό στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας αλλά ούτε και η Επιτροπή υπερεύει αυτή την αρχή που όλοι τη συμμεριζόμαστε αυτή της επικορικότητας και εγώ συμφωνώ μαζί της το μοναδικό σχετικά με τις οδηγίες για κανονισμούς δεν έχουν να κάνουν με νέες οδηγίες, νέους κανονισμούς που σαν εισηγητής εγώ επιθυμώ να συμπεριλάβει κάτι το καινούργιο το κοινό κανείς ε, δεν επιθυμώ κάτι τέτοιο. Το μοναδικό είναι ε, οι υπάρχουσες οδηγίες, υπάρχοντες κανονισμοί που θα πρέπει κάπως να επικυροποιηθούν ή να συζητηθούν ε, και η οδηγία για τα ταξίδια υπάρχει ήδη και πολλές, σε πολλές συζητήσεις είπαμε ότι θα πρέπει να το ανανεώσουμε τον Ατάλο. Υπάρχει ήδη αυτή η οδηγία, θα πρέπει να τη βελτιώσουμε. Δεν πρόκειται για καινούρια δική μου επινόηση. Και ακόμη κάτι για θα περιφορολογικών. Δεν είναι κατομιστικό ότι εργάζονται για το ΦΠΑ υπηρεσίες. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται ε, ο τουρισμός, ε, πώς θα συμπεριληφθεί στη σχετική συζήτηση αλλά κάπως έσπασε αυτό το ταμπού εδώ και αρκετά χρόνια. Τα κράτη-μέλη, τα ε, ευρωπαϊκά όργανα μιλάνε για τα φορολογικά και ε, ε, σταμάτησε αυτό. Εδώ φαίνεται κάτι το παράδοξο όμως. Όταν μιλάμε για την ποιότητα και την ασφάλεια, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι ενώσει καταναλωτών και τα συνδικάτα μας λένε θα πρέπει να έχουμε μια οδηγία, μια ρύθμιση ευρωπαϊκή, ώστε παντού, στο βορρά και στο νότο, ανατολή και δύση της Ευρώπης, θα πρέπει ας πούμε αντιπυρική προστασία να ισχύουν τα ίδια παντού με μια ενιαία ρύθμιση. Βλέπετε ότι εδώ το τονίζω, αλλά να ενταχθεί κάποιος θεληματικά, εθελοντικά και ε, εντάξει με κοινά κριτήρια αλλά ποτέ δεν υποστηρίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια νέα οδηγία, ένας νέος κανονισμός ε, που θα πρέπει να ρυθμίσει ε, ξανά η Ευρώπη, κάτι που έχει ήδη ρυθμιστεί. Εγώ κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια να μην μπω όπως σας είπα σε ξένα χωράφια όπως αυτό της επικουρικότητας και η συνθήκη μας λέει ότι μπορούμε να υιοθετήσουμε μέτρα όμως συντονισμού. Ορισμένα άλλα πράγματα τάχιστα οι επαφές, οι σχέσεις, οι διαπεριφερειακές, ο τουρισμός σαν ε, παράγοντας ε, ανάπτυξης. Οι Σνάφη Δανέλης και Ούγιας το τόνισαν αυτό και εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί τους. Ε, ορισμένα στοιχεία έχω βάλει λίγο μέσα, αλλά από δική σου πλευρά αν θέλουν να προσθέσουν κάτι δεν θα αντιμετωπίσω καμία δυσκολία να τα δοθετήσω κι εγώ. Κάτι ακόμα από αυτές τις παρεμβάσεις σχετικά με το να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες με ειδικέ ημερομηνίε και να προσκαλέσουμε την Επιτροπή την Ευρωπαϊκή να λάβει μέτρα ας πούμε μέσα σε τόσο χρονικό διάστημα. Εγώ και κάποια διαθεσούλα να υιοθετήσω αυτή τη στάση. Σας το λέω ανοιχτά, καθαρά. Εδώ θα πρέπει να δούμε το όμως ότι δεν υπάρχει και προσωπικό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έχουμε μία μονάδα, ένα τομέα τουρισμού. Υπάρχουν άξιοι, πανάξιοι υπάλληλοι, αλλά από προσωπικό δεν υπάρχει και πολύ. Λίγοι και καλοί, αλλά όχι πολυ Άρα λοιπόν, ε, γι' αυτό θα πρέπει να δούμε αυτές τις προτεραιότητες. Ε, θα πρέπει να δούμε μια συνεχή επαφή με την Επιτροπή την Ευρωπαϊκή, χωρίς να τους επιβάλλουμε, ας πούμε, σε τρεις-έξι μήνες, ένα χρόνο τους επιβάλλουμε αυτό, γιατί όλα αυτά... Ε, έχουν άμεση σχέση με τη δυνατότητα πλευράς Επιτροπής να κινητοποιήσει κόσμο προσωπικό για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Τώρα πλευρά αδέλφου Βρέπος που είπε ότι ε, ένας κανονισμός για την προστασία των τουρισμών, εντάξει, το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε και είδαμε τους διάφορους κανονισμούς για τους ε, επιβάτες, για τους τουρίστες, την προστασία τους. Εμείς σαν Επιτροπή εδώ οθούμε προς ένα νέο κείμενο που να συμπεριλαμβάνονται όλοι οι κανισμοί αλλά τώρα ε, φοβάμαι να ξεκινήσουμε ειδικού ειδικού ε, ε, κανόνες, κανονισμούς για τους τουρίστες. Έχουμε ε, ε, τύχη καλύψω άρρωστε που θα πρέπει να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά. Και πετούνται βέβαια και χρήματα, κονδύλια, αλλά ήδη το καλυψό έδειξε δυνατότητες και να δούμε και τους υλοκιωμένους συνταξιούχους κλπ. Αυτό σίγουρα θα πρέπει να υποστηριχθεί. Σταφος Μπακ για το Digital Plus κλπ. Εδώ υπάρχει ήδη αυτή η δράση και η οποία συμπεριλαμβάνεται στο Small Business Act. Αναφέρεται δε σε τρεις τομείς οι οποίοι έχουν να κάνουν με τη μόδα, τα υφάσματα, μεταφορά, οργάνωση και με τα ε, αυτοκίνητα θα πρέπει να δούμε πώς θα διευρυνθεί η εφαρμογή αυτής της δράσης, αυτού του προγράμματος και στην τουριστική βιομηχανία. Ένα τελευταίο θέμα τώρα για την πρόσβαση και για τις μεταφορές και στο λέω ειλικρινά, ειλικρινά. Εδώ η έκθεση αυτή που έχει να κάνει με τον τουρισμό και τις μεταφορές ίσως θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο. Ανέφερα σε περιπτώσεις με δηλώσεις αρχών και απόψεων, αλλά τα μέλη εδώ ίσως θα μπορούσαμε να εμπλουτίσουμε, να κάνουμε αποτελεσματικότερο το κείμενο αυτό και για την πρόσβαση σε πιο δύσκολες για πρόσβαση περιοχές. Άρα λοιπόν είμαι έτοιμος να ακούσω και υποδείξεις πάνω σε αυτά τα θέματα και σας ευχαριστώ όλους σας για τη συνεργασία σας. 8 Μαρτίου είναι η προθεσμία. Επίσης, θα γίνει εξέταση στον Απρίλιο. και θα περάσει από την Ολομέλη τον Ιούνιο ή Ιούλιο. Αλλά η τροπολογία τροπολογια ειναι στις 8 Μαρτίου παρακαλώ. Λαμπρά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερχόμεθα τώρα στην υπέρμενη, σε επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης. Κύριε Μπρέμπος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ήθελα να πω κάτι, γιατί στις 8 Μαρτίου, όπως γνωρίζετε, είναι η πρώτη μέρη που θα είμαστε στο Στρασβούργο, 8 Μαρτίου. Είπατε λοιπόν ότι είναι η τελευταία μέρα για τις τροπολογίες. Αυτή τη βδομάδα λοιπόν Είμαστε στην εβδομάδα της εξωτερικών υποθέσεων και αυτή την εβδομάδα έχουμε πάρα πολύ σημαντικές συναντήσεις στη Ρώμη με τους ε, εκπροσώπους της μεσογειακών χωρών και εγώ φεύγω. Ε, αυτός ο λόγος είναι για τον οποίο δεν μπορώ να περιμένω μήπως θα μπορέσουμε να το παρατηρούμε μέχρι τέλος ε, του Στρασβούρου, της Ολομερίας του Στρασβούρου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, για να έχουμε πιο πολύ χώρο, χρόνο. Αν συμφωνούμε, πραγματικά μπορώ να το παρατείνω μέχρι τις 10 του Μαρτίου, μέχρι την 5η 10, δηλαδή μέχρι το πέρας της Ολομελίας του Στρασβούργου. Το πρόβλημα είναι η μεταφράση. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο πραγματικά βιαζόμαστε. Γιατί θα πρέπει να μείνουμε εντός του χρονοδιαγράμματα. Εις 12, ε, τώρα ήταν 10 λέει. 10. Συμφωνείτε ησυχητά. Ωραία, Λάμπρα, σας δίνω μέχρι τη δεκάτη Μαρτίου. Μαρτίου. 10 Μαρτίου, συνεπώς. Επόμενο σημείο της μέρης διάταξη είναι οι στατιστικές όσον αφορά στον τομέα του τουρισμού και θα ήθελα να δώσουμε τις ευκαιρίες για να σας πω ότι θα πρέπει να επανέλθουμε την περιεπιτροπή όσον αφορά τη διαβάθμιση που πρέπει να γίνει με το Συμβούλιο και για να υπάρχουν ε, το πλαίσιο εκείνο το οποίο θα είναι χρήσιμο για τη συλλογή των στοιχείων στερεοφορώτων τουρισμού. Υπάρχουν ανεπίσημες επαφές αυτή τη στιγμή με την Υπηρετική Προεδρία και στο τέλος χρονιάς ξεκίνησε ένας τρίλογος, τρι, τριμερής διάλογος και υπήρξε μια πρώτη ανάγνωση στην οποία συμφωνήθηκε και θα ήθελα να ευχαριστώ τον κ. Φουντάτσα, κ. Ντουράν επίσης οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την, τον τριπλό διάλογο όταν έλαβε χώρα. Ε, φρονώ λοιπόν πως το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό. 22-20 ε, τροπολογίες έγιναν, από τις 29 έγιναν ε, αποδεκτές στο κείμενο και περιλαμβάνει τα οποία, αυτά τα οποία επιβάλλουν περιορισμούς στην Κομισιόν όσον αφορά βεβαίως τον ορισμό αυτή της, κατά αυτής της υπόθεσης και βεβαίω αυτά μπήκαν στην όλη διαδικασία. Ιδιαίτερα θα ήθελα να πω για το παράρτημα το οποίο βάζει πολλές στατιστικά στοιχεία και τα οποία ε, βεβαίω είναι πολύ χρήσιμα. Συμφωνήσαμε όλοι λοιπόν αυτή τη στιγμή να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη ε, πιλωτικές εργασίες όσον αφορά τον τουρισμό και επίσης πώς πραγματικά συμβάλλει στην οικονομία, στην απασχόληση και δεχτήκαμε τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η οποία δέχτηκε αυτή τη στιγμή τις πιλωτικές εκείνες στατιστικές ομάδες που θα επιδεικνύουν τον τουρισμό και την επίπτωση του τουρισμού στο επιπεριβάλλοντος. Άλλες τροπολογίες οι οποίες ελήφθαν υπόψη είναι η τροποποίηση του κανονισμού και τα παραστήματα που εισήχθησαν αυτοί καθώς επίσης και στα οποία περιλαμβάνονται ακόμη και τα έξοδα των εστιατορίων. Υπάρχει λοιπόν ε, ένας ορισμός σαν αφορά την ε, ημερήσια εκδρομή και τον κοινωνικό τουρισμό, ε, κοινωνικό τουρισμό συγγνώμη, επίσης. Επίσης θα επιβεβαιωθούν, επιβεβαιώθηκαν αυτά τα στοιχεία της συνάντησης της 1 Φεβρουαρίου και τα, οι βουλευτές θα βρουν αυτή τη στιγμή μέσα στο φάκελό τους τα αντίστοιχα κείμενα. Επίσης τα μόνα θέματα τα οποία μένουν εκρεμές είναι, είναι περίληψη των στατιστικών όσον αφορά την προσβασιμότητα ε, για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ελαττωμένη κινητικότητα. Νομίζω πως δεν συμφωνήσαμε σε αυτό το σημείο για τη διατύπωση που θα έπρεπε να γίνει. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή εγώ, υπάρχουν συζητήσει ακόμη αυτή τη στιγμή με το Συμβούλιο για αυτό το θέμα και πιστεύουμε ότι έχει γίνει κάποια πρόοδο στη τελευταία συνάντηση του Συμβουλίου στις 25 Φεβρουαρίου. Δεν έχουμε τίποτα αυτή τη στιγμή, τίποτα επίσημο το οποίο εξεδόθηκε εκ, εκ του μέρου του Συμβουλίου, αλλά πιστεύω πω πραγματικά θα συμφωνήσει τελικά σε αυτό το θέμα, σε αυτή την προσβασιμότητα των ανθρώπων με αναπηρίε, με μειωμένη, αν θέλετε, κινητικότητα. Και δεν μπορώ να είμαι αυτή τη στιγμή, αλλά περιμένω επιβεβαίωση εκ μέρου του Συμβουλίου μετά την συνάντηση 25 Φεβρουαρίου. Αυτό, εάν συμβεί πραγματικά, τότε εγώ φρονώ πως η συμφωνία θα είναι μια μεγάλη επιτυχία για το Κοινοβούλιο και πραγματικά εφόσον το έχουμε αυτή τη στιγμή και το πετύχουμε όλο αυτό και όλα αυτά που πετύχαμε νομίζω πως πραγματικά θα υπάρχει ένα κείμενο μόλις τροπολογίες που έχουμε και το που έχουμε εισάγει καθώς επίσης και τις ελαφρές εκείνες αλλαγές οι οποίες έχουμε εισαγγελία για την εφαρμογή του. Επίσης θα πρέπει ε, να επιβεβαι... αρχές Μαρτίου αυτό το κείμενο και πιστεύω πως θα περάσει στην Ολομέλεια του Μαρτίου Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις βέβαια αυτή τη στιγμή, η συμφωνία μπορεί να έχει συμφωνηθεί τελειωτικά και να μπει η τελική σφραγίδα με αυτή τη βάση. Εγώ λοιπόν επαναλαμβάνω ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχή με αυτό το κείμενο και την εργασία η οποία έχει επιτελεστεί ιδιαίτερα σε αυτό τον τριπλό διάλογο που έχει γίνει, τριμερή διάλογο συγγνώμη, και νομίζω πως πραγματικά είναι ένας τρόπος με τον οποίο δρούμε εμείς αυτή τη στιγμή και χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή την επιβεβαίωση, διότι έτσι έχουν τα πράγματα και έτσι προχωρούν τα πράγματα. Κύριε Φιδάνιτζα, έχετε το λόγο παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν θα ήθελα να προσθέσω σχεδόν τίποτα σε αυτό που είπατε εσείς. Είπαμε μαζί ποιες ήταν οι προτεραιότητες της διαπραγμάτευσης με το Συμβούλιο. Νομίζω ότι καλύτερο και από αποδεκτό σκέτα είναι το αποτέλεσμα και περιορίσαμε το θέμα στα μην ε, απαραίτητα μέρη και αφήσαμε και τα υπόλοιπα στην πλαίσια της τακτικής διαδικασίας επίσης στη μελέτη πιλότ για τους υπόλοιπους ε, βοηθητικού λογαριασμού και επίσης οι ημερήσιες επισκέψεις χάρη στην εργασία μας εντάχθηκε και αυτό στο, σε ένα σωστότερο πλαίσιο, διευκρινίστηκε καλύτερα στο κείμενο αυτό, παραμένει το θέμα για τα άτομα περισμένης κινητικότητας ε, και μετά από τα όσα λίγα μας είπα την τελευταία συνάντηση στην ομάδα εργασίας δεν ξέρω νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να επιβεβαιωθούν ακριβώς ώστε να έχουμε και αυτή την προτεραιότητα της Επιτροπής μας ε, αυτό που υποστηρίζουμε να γίνει δεκτό και να προβληθεί και από το Συμβούλιο. Υποστηρίζουμε λοιπόν αυτή τη θέση και ελπίζουμε τα πράγματα να πάνε προς την κατεύθυνση αυτή κύριε Στέιλορ, παρακαλώ, έχει το λόγο. Πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να μην χάσω την ευκαιρία αυτή τη στιγμή, χωρί να πω το εξή. Ότι εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, νομίζω πω πραγματικά αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε με το. Πρέπει να δοθεί αυτή η δυνατότητα με του ανθρώπου που έχουν μειωμένη προσβασιμότητα και νομίζω πραγματικά ότι ενθερνόμεθα όλοι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και παρακαλώ πρόεδρε να επιμείνετε για αυτό το θέμα. Ναι. ναι, Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, βέβαια δεν το πετύχαμε όλα, αλλά ναι. Ο κύριος Ντιμόντα έχει παρακαλώ το λόγο εκ μέρους της Κομισιόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σιγητά. Συμφωνώ απόλυτα ότι, ότι πραγματικά ήταν πάρα πολύ κοινοποιητική και όλα τα μέρη σε αυτόν τον τριήμερη διάλογο το οποίο έχει γίνει επέτυχαν πέτυχαν του σκοπούς τους. Έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο παραμένει αυτή τη στιγμή σε κρεμότητα όσον αφορά τα άτομα με ελαττωμένη προσβασιμότητα και κινητικότητα, συγγνώμη, και μου φαίνεται πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο, το οποίο δεν μπορεί να το διαπραγματευτεί να υποχωρήσει το Κοινοβούλιο από αυτό το θέμα, όπω καταλαβαίνετε. Για να διορθώσω κάτι αυτή τη στιγμή, δεν υπήρχε 25η ε, Φεβρουαρίου ε, συνάντηση. Απλούστατη η Προεδρία ότι συνήλθε με τη συναντήση και δεν ελήφθη βέβαια το θέμα αυτό ε, απλούστατα την, την προηγούμενη Παρασκευή εδέχθηκα μόλις τρεις μέρες πριν εδεχθήκαμε πραγματικά την απάντηση των κρατών μελών όσον αφορά το θέμα αυτό το οποίο έχει και βεβαίω θα πραγματικά πάνω στα ξενοδοχεία, σε άλλα τα θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα πρόσβαση των ανθρώπων με προβλήματα κινητικότητα. Εμεί επίση κοιτάζουμε ε, να δούμε μπροστά, βλέπουμε προς τα μπρος για να δούμε πραγματικά ποια θα είναι η απάντηση η οποία θα δοθεί και πώς θα επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα το οποίο ανακύπτει για αυτά τα άτομα. Υπάρχει μια μεταβατική περίοδο και ε, η οποία θα ξεκινήσει μέσα από την Επιτροπολογία η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή σε αυτό το θέμα και βεβαίως θα έρθει στην Επιτροπή προς ψήφιση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, Περιμένουμε να δούμε πραγματικά το Συμβούλιο τι θα γίνει, πώς θα το εξετάσει και πώς θα το ε, περατώσει αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Λαμπρά. Ευχαριστώ. Το επόμενο σημείο της ημερήσια διάταξη Κόχ έκθεση ε, Ευρωπαϊκή Οδική Ασφάλεια Δίτερ, θα ήθελες να παρουσιάσεις την έκθεση σου παρακαλά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, τι θα ήταν ο τουρισμός χωρίς την κινητικότητα. Αδιανόητο θα ήταν. Και τι θα ήταν η κινητικότητα χωρίς ασφάλεια. Και πάλι αδιανόητο. Γι' αυτό πιστεύω ότι ταιριάζουν πολύ μεταξύ τους οι εκθέσεις τις οποίες συζητάμε σήμερα. Με την δική μου έκθεση θέλω να μιλήσω για την Ευρωπαϊκή Οδική Ασφάλεια από το 2011 μέχρι το 2020. Θέμα ιδιαίτερα σημαντικό και όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να δημιουργήσουμε κίνητρα ε, σε όλα τα επίπεδα, σε εθνικό, σε περιφερειακό, τοπικό επίπεδο, γιατί η κινητικότητα που είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα θέλουμε να γίνει ακόμη ασφαλέστερη και για όλους αυτούς που συμμετέχουν στις μεταφορές και για τους πεζούς και για αυτούς που μετακινούνται με αναπηρικά καροτσάκια και για τους ε, επιβάτες οχημάτων και Γι' αυτό στην έκθεσή μου τονίζω ιδιαίτερα το τρίτο πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οδική ασφάλεια. Όχι όπως στην έκθεση πέντε στην προηγούμενη θητεία, γιατί αυτό το οποίο έγινε ε, τότε νομίζω ότι έχει περιπέσει σε λύθη πλέον. Υπάρχουν ε, διαφορετικοί τομεί αρμοδιότητα. Για κάποιου τομεί ε, είναι αρμόδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, για άλλου τομεί ε, τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο ή περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο με τι αντίστοιχε αρχέ αυτοδιοίκηση και πολύ συχνά είναι, έχουν αρμοδιότητα οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι στι μεταφορέ, οι ίδιοι οι οι πολίτες. Ε, οι πολίτες ε, έχουν και δικαίωμα στην πληροφόρηση, αλλά έχουν και, δικαίωμα, έχουν και υποχρέωση συμμετοχής. Και θέλω να τονίζω ότι εμείς αναλαμβάνουμε ευθύνη για τον εαυτό μας και για τους άλλους όταν συμμετέχουμε στις μεταφορές, με ή χωρίς όχημα και πολύ συχνά είμαστε παρατηρητές του ότι οι πολίτες δεν έχουν επίγνωση των ευθυνών τους. Δεύτερον, ε, είναι μεγάλη πρόκληση γιατί ε, ήδη τα προηγούμενα χρόνια έχουμε επιτύχει πάρα πολλά. Την περασμένη Παρασκευή στη Γερμανία άκουσα στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο μια αξιολόγηση σχετικά με τον αριθμό των ατυχημάτων και τον αριθμό των θυμάτων ε, και φαίνεται ότι από τότε που αρχίσαμε να κρατάμε στατιστικά στοιχεία έχουν μειωθεί τα θύματα και είχαμε τον, ε, ε, με την τελευταία καταμέτρηση το μικρότερο αριθμό θυμάτων και γι' αυτό είναι και πιο δύσκολο να επιτύχουμε περαιτέρω μειώσεις των αριθμών ατυχημάτων και θυμάτων. θα ήταν καλό όλοι να έχουν επίγνωση και να τηρούν ε, τις αντίστοιχες ε, διατάξεις. Θα έπρεπε να έχουμε επίγνωση του κινδύνου όταν μπλεκόμεθα στις μεταφορές και όταν ε, εμείς παίρνουμε μέρος στις μεταφορές θα πρέπει να γνωρίζουμε τον κίνδυνο το οποίο διατρέχουμε εμείς και διατρέχουν και οι άλλοι αν δεν είμαστε υγιείς ή αν δεν είμαστε σε κατάλληλες ε, συνθήκες. Παράλληλα θα πρέπει να παραμείνουμε πρακτικοί και ρεαλιστές. Υπάρχει η ε, μηδενική προοπτική, το Vision Zero δηλαδή, με μηδενικό αριθμό ατυχημάτων ως στόχο θα πρέπει να προσπαθήσουμε ε, να τηρήσουμε ε, στο μέτρο του δυνατού αυτά τα οποία ε, προτείνονται. Για να έχουμε μηδενικό αριθμό ατυχημάτων θα χρειαζόμασταν υπερβολικά υψηλό επίπεδο πόρων και θα χρειαζόμασταν ε, δέσμευση πόρων ε, που θα ήταν ε, υπερβολικά υψηλή σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους και νομίζω ότι δεν θα ήταν κατάλληλο, κατάλληλο στόχος. Πιστεύω ότι θα υπήρχαν μειονεκτήματα και για την κινητικότητα των πολιτών και για την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Θέλουμε λοιπόν να βελτιώσουμε την οδική ασφάλεια με υπευθυνότητα και με συνολική θέαση των επιπτώσεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και ιδιαίτερα τους δυο συζητητές για τις πολλές ε, παρατηρήσεις και σχόλια που μου έκαναν που σίγουρα δεν πήγαν χαμένα. Προσπάθησα να τα συμπεριλάβω όλα στην έκθεσή μου. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τη γραμματεία της Επιτροπής μας, ε, Dan Clefson, για την κυρία Γκράουελ για την υποστήριξή τους και για την ε, συστηματοποίηση των πολλών προτάσεων που υπευλήθησαν κατά τη διαμόρφωση της έκθεσής μου. και θέλουμε να υποστηρίξουμε αυτά τα οποία γίνονται σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο και τονίζουμε και τα βασικά σημεία της έκθεσής μου. Στην έκθεσή μου καταρχήν ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω την έκθεση αυτή, ούτω ώστε να καταλήξουμε σε ένα πρόγραμμα δράσης μέχρι το 2020 για την οδική ασφάλεια και προτείνω η Επιτροπή μέχρι τα τέλη του έτους να έχει υποβάλει μια σχετική πρόταση. Μιλάμε για ασφαλή και καθαρή κινητικότητα σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ χρειάζεται σαφώς συντονισμός μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη πιστεύω ότι η πολυπλοκότητα των απαραίτητων ε, μέτρων που ε, πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη, αλλά και οι επιχειρήσεις ε, και όλοι όσοι συμμετέχουν στις μεταφορές, χρειάζονται συντονισμό. Και γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργηθεί μια θέση συντονιστού για τις οδικές μεταφορές ε, τρίτον, υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα τα οποία θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά. Θέλουμε να μειώσουμε βεβαίως τον αριθμό των ε, τροχαίων ατυχημάτων και ιδιαίτερα των θανατηφόρων ατυχημάτων. Ε, εδώ νομίζω ότι είναι σημαντικό το να έχουμε και ενιαίους ορισμούς και συγκρίσιμα στατιστικά δεδομένα. Βέβαια, υπό την ε, τη φύλαξη ε, της διαφύλαξης ε, και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αλλά θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά τα στατιστικά δεδομένα. Την επιδίωξη του μηδενικού αριθμού ατυχημάτων ε, μπορεί να μην τη θέσουμε ως στόχο για το 2020 αλλά αυτό το Vision Zero δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε ως ε, απότερο στόχο μας. Ακόμη θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό και τους οδηγούς ε, και τους, όλους τους πολίτες που συμμετέχουν στις μεταφορές και στην κινητικότητα μέτρα ευαισθητοποίησης με εκστρατείες ενημέρωσης και άλλους τρόπους. Στην περαιτέρω εναρμόνιση και ε, τήρηση των διατάξεων για την οδική ασφάλεια στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς οδικής ασφάλειας θα πρέπει να προωθήσουμε όλα αυτά τα μέτρα. Γιατί όταν θέλουμε να έχουμε πιο ασφαλείς οδικές υποδομές και θα πρέπει να τηρούνται οι ισχύουσες προδιαγραφές ούτως ώστε να χρηματοδοτούνται ε, οι υποδομές αυτές. τα οχήματα, τέταρτον, τα οχήματα θα πρέπει ε, να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ε, ασφάλειας και σε σχέση με τις νέες μεθόδους κίνησης των οχημάτων, παραδείγματος χάρη ηλεκτρικά οχήματα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη νέες τεχνολογίες, καθώς ε, και η προμήθεια εξαρτημάτων και ανταλλακτικών Πέμπτον, θέλουμε νέες τεχνολογίες να ισχύσουν για τα οχήματα, αλλά και για τις υποδομές ε, παροχής ε, υπηρεσιών και ε, υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, παραδείγματος χάρη. Στα ευφυή e συστήματα μεταφορών χρειαζόμαστε και ευφυή e συστήματα οδικής ασφάλειας για την αποφυγή των ατυχημάτων ή για την ελαχιστοποίηση του αριθμού των ατυχημάτων και παράλληλα υποστήριξη από υπηρεσίες ε, παροχής πρώτων βοηθειών ε, στο κατάλληλο επίπεδο θέλουμε να, ισχύει οδική ασφάλεια για όλους τους ε, συμμετέχοντες στις μεταφορές και ιδιαίτερα για τους ποδηλάτες, τους μοτοσυκλετιστές, τους πεζούς, ε, τα παιδιά. Προσπάθησα να περιορίσω τα σχόλιά μου σε αυτά τα οποία είχα τη δυνατότητα μέσα στον αριθμό των λέξεων που μου επιτρέπετε ε, και θα ήθελα με τις δικές σας τροπολογίες να συμπληρώσετε αυτά τα οποία εγώ ενδεχομένως έχω παραλείψει και να συνεχίσουμε την ε, επικοδομητική συνεργασία μας. Υπάρχουν ε, διάφορες προτάσεις, ε, προτάσεις για τα 5 λεκ που είναι τα ποδήλατα με ηλεκτρική υποβοήθηση, προτάσεις για τις εκστρατείες που μπορούν να γίνουν για την ε, οδική ασφάλεια, ενδεχομένως προτάσεις για κάποιες πιλωτικές περιοχές, ούτως ώστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο για την οδική ασφάλεια. Σας ευχαριστώ πολύ και θα περιμένω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε εκτιμώ πάρα πραγματικά και ξέρω ποιες δυσκολίες υπάρχουν όταν πραγματικά αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η δυσκολία όσον αφορά και την κατάσταση. για yeah, συγγνώμη αυτή τη στιγμή ε, εκτιμώ ότι αυτή τη στιγμή και η δική σας και του κ. Φιντάντζα η εκθέση είναι συγγνώμη που το λέω αυτό το πράγμα αλλά είναι ε, είμαι υποχρεωμένος να το πω ότι είναι δύο εκθέσεις οι οποίες πραγματικά ε, προωθούν τη δική μας δουλειά κύριος Αρκατράουι, ο οποίος είναι σκιώδης αυτή τη στιγμή. Τρία με τέσσερα λεπτά μάξιμα παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρόεδρε. Ε, εγώ θα μιλήσω ο Στεφανίων, ο οποίο που δεν μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω για την προσέγγιση του τον εισηγητή και είναι μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση και συμφωνώ μαζί του. Νομίζω πω άπτεται όλων ημών και νομίζω πως καλέ καλές σωστέ πολιτικέ θα μπορούν να, μπορούν να προλάβουν πάρα πολλού θανάτου κάθε χρόνο. Και αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο είναι πάρα πολύ σημαντική η έκθεσή σα. Επίση, είναι και καλή ευκαιρία να σκεφτεί κανένα τι θα πρέπει να επιληθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πώς θα πρέπει να ρυθμιστεί και άλλοι όχι. Ε, ελέγχθηκαν πολλές πραγματικά αυτή τη στιγμή προτάσεις ε, για, για τους τροχούς κλπ. Η κατάσταση είναι τόσο διαφορετική από τις άλλες χώρες που δεν ξέρω πραγματικά. Υπερκέρ, Υπάρχουν περιοχέ οι οποίε είναι πάρα πολύ με υπερπληθυσμό, άλλε είναι με λιγότερο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε αυτή τη στιγμή ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση που μπορούμε να έχουμε σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν όμω πολλέ περιοχέ όπου πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν ευρωπαϊκά μέτρα τα οποία θα, θα καλύπτουν αυτέ τι περιοχέ. και νομίζω πω αυτό είναι μια εξαιρετική ιδέα η οποία ξεκίνησε ότι θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να λεφθούν μέτρα. Μη είπατε για αυτού τους αλκοολόγους ε, συστήματα κρυδόμως των αρκολόγων και πως αυτό πραγματικά νομίζω πως πραγματικά αυτό ισχύει όσον αφορά το φορτηγά ήδη έτσι και πάει καιρό αυτό το οποίο υπάρχει εδώ όταν μιλάμε για αυτή τη στιγμή για το θέμα του διοξιδίου του άνθρακος και της πώς πραγματικά ε, ξέρετε αυτό το θέμα όσον αφορά το διοξείδιο του άνθρακος έχει περάσει από την Ολομέλεια ή ε, θα πρέπει να δούμε αυτά τα μέτρα ξανά και κατά πόσο πετύχουμε κάτι περισσότερο όσον αφορά τον περιορισμό της ταχύτητας οποία υπάρχουν και πρακτικά πράγματα τα μετρα ξανα και τα ποσο ανακύπτουν πολλά προβλήματα τα οποία κοινοτική αυτή τη στιγμή ε, ευχαριστώ φοβερά θέματα τα οποία πραγματικά είναι μια σειρά ολόκληρα θέματα τα οποία θα πρέπει να τα ρυθμίσουμε και τα οποία άπτονται τη δική μα αρμοδιότητα αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή βάση των σαρβατών ο, ο ορισμό που θα πρέπει να υπάρχει αυτό. Νομίζω πως πραγματικά πρέπει να υπάρχει ένας συντονιστής όσον αφορά την εωδική ασφάλεια. Δεν είναι μια καλή ιδέα αυτή το πράγμα. Και θα πρέπει να είναι μέσα στην Επιτροπή. Πώς πραγματικά πώς μπορεί η Γενική Διεύθυνση μπορεί να κινηθεί σε αυτό το θέμα στα πλαίσια της Κομισιόν και πώς μπορούμε να βρούμε μία λύση και πώς πραγματικά μπορούμε να βασιστούμε σε κάτι μέλη, ναι, μέλη, ναι ή όχι. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός συντονιστής για αυτό το πράγμα, ευρωπαίος συντονιστής, συγγνώμη. Επίσης η κατάρτιση πιστεύω πως μπορει η γενικη διευθυνση μπορει να κινηθει σε αυτο το θεμα στα πλαισια της κομισιον και πως μπορουμε να βρουμε μια λυση και πως πραγματικα μπορουμε να βασιστουμε σε κατι μελη ναι ναι η οχι εν παση περιπτωσει θα πρεπει να υπαρχει ενας ευρωπαικος συντονιστης για αυτο το πραγμα ευρωπαιος συντονιστης συγγνωμη επισης η καταρτιση πιστευω πως πραγματικη ε, σε αυτό το σημείο επίσης μπορεί να υπάρξουν οδηγίες καθώς επίσης και κατηγορίες, τα παιδιά, τα δίκυκλα, τα ποδήλατα κλπ. 14 ετών είπατε, δεν θα πρέπει πραγματικά αυτό να ισχύει για όλα τα παιδιά, άσχετα είναι 14 ή όχι. Επίσης για τα οχήματα πρέπει να δούμε νέες καινοτομίες, ηλεκτρικά αυτοκίνητα κλπ. Και επίση θα πρέπει να υπάρχει μια έξυπνη μεταφορά, ένας μηχανισμός μεταφορά, καθώς επίσης και καινοτομίες. Δεν είναι μόνο τα ηλεκτρικά, αλλά γενικότερα η καινομία η οποία θα πρέπει να υπάρξει σε αυτό το θέμα. Επόμενος, η επόμενη αγόρηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω πριν από οτιδήποτε άλλο τον κύριο εισηγητή για την εξαιρετική έκθεσή του, ότι μας άκουσε για τις καλές σχέσεις τις οποίες έχουμε διατηρήσει κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της προετοιμασίας και να του πούμε απεικόμε ότι καταλαβαίνω πάρα πολύ την απογοητευσή του ότι δεν μπόρεσε μέχρι τούδε να βάλει όλα τα στοιχεία και να τα εξηγήσει μας στην έκθεση που έχει, στο πρώτο, στο πρώτο κείμενο. Δεν θα επανέλθω λοιπόν σε αυτά τα οποία ελέγχθησαν μέχρι τούδε και ασπάζουμε, ιδιαίτερα την έννοια που πρέπει να έχουμε για να επιτύχουμε να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο που είναι πάρα πραγματικός υψηλός στόχος ότι τα άτομα θα πρέπει να μειωθούν κατά το ίμιση οι πεθαίνουν οι δολοφονούμενοι καθώς στην οδική, στις οδικές αρτηρίες καθώς και οι τραυματίες. Και βεβαίω μέχρι τούτο όλα αυτά τα πράγματα ήταν τι δεκακή στο ευρωπαϊκό ε, επίπεδο τη νομοθεσία αναφορά. Έτσι λοιπόν συμφωνώ απολύτω για τη σημασία την οποία έχει και ο συνάδελφό μας δίνει ιδιαίτερα θέμα στην κατάρτιση και την εκπαίδευση σε μια Ευρώπη η οποία γερνάει όλο και περισσότερο καθώς επίσης και στις προτάσεις οι οποίες υπάρχουν να φανταστούμε πώς μπορούμε να λάβουμε υπόψη από τα νιάτα και την εφηβεία την κατάρτιση των νέων 14 ετών για παράδειγμα από 14 και λοιπά να υπάρχει μια συνείδηση οδική επίσης ασπάζουμε την ιδέα ότι χρειάζεται να υπάρχει μια εργασία η οποία θα είναι βαθύτερη για την βελτίωση των οδικών αρτηριών. Υπάρχουν μερικά σημεία, μια και έχουμε λίγο χρόνο, θα πάω στα σημεία τα οποία είναι τα πιο σημαντικά κατ' εμέ και τα οποία θα έπρεπε να εμβαθυνθούν ή να φανούν πιο ισχυρά. Το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση των κυρώσεων. Εάν εξαρ... αυτό εξαρτάται από την κυκλοφορία είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά βέβαια είναι και καλό, αλλά και υπεραπαραίτητο αυτή τη στιγμή Μέχρι στιγμή υπάρχει μία άμεση αναφορά παραπομπή η οποία γίνεται όσον αφορά την αναρμόνιση των κυρώσεων όσον αφορά τις παραβάσεις. Εφόσον δεν υπάρχουν κυρώσεις οι οποίες θα είναι εναρμονισμένες ε, κατά την άποψή μου δεν μπορούμε πραγματικά να βελτιώσουμε την ασφάλεια καθότι υπάρχει μια αίσθηση του ε, ε, έλλειψη ποινών και έλλειψη ε, κυρώσεων σε αυτό το θέμα. Αυτό είναι όλο και το οποίο το προηγούμενο Δεκέμβριο. Εγώ υπο, υποστηρίζω αυτό το οποίο έρχεται όσον αφορά τι διακρατικέ κυρώσει οι οποίε θα πρέπει να υπάρχουν. Δεύτερο σημείο το οποίο είναι στα πλαίσια πάνω τη εναρμόνιση και είναι από τι βασικέ αρχέ τη ΕΕ, νομίζω πω θα πρέπει να εργαστούμε και θα πρέπει αυτή την έκθεση να την ξεκινήσουμε σαν μια απαρχή της όλης προσπάθειας για μια καλύτερη οργάνωση μιας ενοποίησης και ομοιομορφοποίησης όσον αφορά του αρωτά ορίου ε, ταχύτητας, διότι δεν είναι normal αυτή τη στιγμή να υπάρχουν τέτοιες μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα και ιδιαίτερα όταν κανείς είναι ε, ναρκωτικών ή υλοπνεύματο. Δεν ξέρω πραγματικά πόσο γίνεται το ποσοστό, αλλά είναι πολύ ψηλό αυτή τη στιγμή. Το, τα ατυχήματα προ, ε, προκαλούνται από αυτούς που έχουν πάρει ναρκωτικά ή ενόπνευμα, έχουν πιει ενόπνευμα. Επίσης θα πρέπει να μειώσουμε πάρα πολύ ακόμα περισσότερο την αλκοολε, ε, αλκοολεμία και ιδιαίτερα όσον αφορά του, σε σχέση με τους νέους, ένα σημείο όσον αφορά την αρμόνιση πάντοτε, την η χρήση της τεχνολογίας για την ασφάλεια των οδών. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό αυτό και γιατί όχι να μην χρησιμοποιηθεί το καλλιλαίο για να συλλέξουμε τις πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες και να δίδονται στε δετε χρόνο και όσον αφορά το θέμα της βοήθειας, της μέρημνας για την ταχύτητα, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή μερικές φορές απορριθμίζονται, διαρωτώμε λοιπόν πώς θα αυτή τη στιγμή να είχαμε δυνατότητα να ε, βάλουμε ε, τέτοιου είδους εγκαταστάσεις που πραγματικά αυτό και αυτόματα να μειώνουν την ταχύτητα. Ε, έχω πολλά να πω αυτή τη στιγμή κύριε Πρόεδρο και για αυτά τα θέματα όσον αφορά το, την την ε, καθώς επίσης και τους μοτοσυκλετιστές αλλά θα επανέλθει το Δημήτρη επί του θέματος εν ευθέτω χρόνο ο κύριος Τέιλερ παρακαλώ έχει το λόγο ευχαριστώ πρόεδρε Πιστεύω πραγματικά αυτή τη στιγμή έχουμε ε, πολλές τροπολογίες και επανέρχομαι σε αυτό το θέμα και νομίζω πως αυτές ε, ε, είναι οι εκτιμήσεις οι οποίες και επανέρχομαι εδώ στις εκτιμήσεις οι οποίες έγινε εκ μέρους του εισηγητού για μια αλλαγή η οποία θα είναι μίζω και πρέπει να γίνει. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα για τα οποία πραγματικά έχω πολύ ισχυρά σημεία τα οποία θα πρέπει να υποβάλω και με τον κύριο Κόκ για παράδειγμα και εκτίμησα τη συνεργασία, τα υπέβαλα και εκτίμησα αυτή τη στιγμή τη δική του. Αλλά όταν στην ουσία πραγματικά κοιτάξω το πράγμα νομίζω πως τα δεν βλέπουμε σωστά. Εδώ είναι μια έκθεση η οποία μιλάει για την αστεοδική ασφάλεια. Το λέω αυτή τη στιγμή και το θέτω γιατί η ασφάλεια οδική είναι ασφάλεια. Δεν έχει σχέση. 35.000 ε, άτομα αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο το αυτό το θέμα, γιατί ο κύριος μας ζήτησε αυτή τη στιγμή κατά πόσο θέλουμε να θέσουμε ε, ε κατά πόσο θέλουμε αυτή τη στιγμή να, να μειώσουμε την, την ορατότητα σε μηδέν. Δεν, νομίζω πως θα πρέπει να έχουμε πολύ περισσότερη φιλοδοξία, αποφασιστικότητα, όραμα και αποφασιστικότητα. Να μην το δεχθούμε αυτό το πράγμα. Είναι ένα σημαντικό θέμα που άπλεται όλη την κοινότητα. Έχει ένα φοβερό ε, επίπτωση αυτή τη στιγμή, δραματική επίπτωση όσον αφορά και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πολύ πιο δυναμικά αυτό το θέμα μέσα σε αυτή την έκθεση. Όταν λοιπόν έρχομαι αυτή τη στιγμή τη τροπολογία τη οποία έχω καταταθεί και όταν λέγω ότι πρέπει να το σκεφτείτε, θέλετε να πείτε αυτή τη στιγμή ε, ότι υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πεθαίνουν και θα, και θα πρέπει αυτό το πράγμα να το δούμε πάλι. Ευχαριστώ κύριο Μπράντμπρουν. Τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κατανοώ τις προσπάθειες ε, του κύριου Κόχ. <coughs> Οφείλω όμως να πω ότι ε, αποδείξετε αυτό που περίμενα και εγώ στο οποίο θα καταλήγαμε με μια τέτοια έκθεση. Ε, όλοι θέλουμε να βελτιώσουμε την οδική ασφάλεια, όλοι είμαστε κατά της αμαρτίας, ε, αλλά πώς θα το κάνουμε. Το θέμα είναι αν υπάρχει κάποιος ρόλος για μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως και άλλοι συνάδελφοι έχουν πει και έχουν ακούσει για το θέμα αυτό, θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα θέμα για τα κράτη-μέλη, για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και όχι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να υποβάλω κάποια σχόλια για συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στην έκθεση του κυρίου Κόχ. Κάποια σημεία αναφέρθηκαν και από άλλους συναδέλφους. Μιλάει για τη διαβίου μάθηση ο κύριος Κόχ. Εγώ οδηγώ αυτοκίνητο πάνω από 40 χρόνια. Κάθε μέρα μαθαίνω. Κάθε φορά που μπαίνω στο αυτοκίνητό μου κάτι μαθαίνω. Δεν χρειάζεται να έρθει κάποιος να μου πει ότι πρέπει να ξανακάνω τεστ οδήγησης μια φορά στο τόσο ε, που είναι ε, γιατί κάτι τέτοιο λέμε στην έκθεση αυτή. Οποιοδήποτε οδηγεί αυτοκίνητο γνωρίζει ότι αλλάζουν οι συνθήκες οδήγησης, ότι αλλάζει η υποδομή και σιγά σιγά προσαρμοζόμαστε. Δεν χρειάζεται κάποιος κανονισμός για να μας κάνει να προσαρμοστούμε σε αυτά που αλλάζουν. Μια άλλη πρόταση τώρα που αναφέρει ο κύριος Κόχ για τα συστήματα κλειδώματο αλκοολόκ. Δεν ξέρω αν προτείνεται να εγκατασταθούν εκ των υστέρων στα οχήματα, ε, αλλά έχετε σκεφτεί πόσο κοστίζουν αυτά. Υπάρχει ένα πολύ καλό τέτοιο σύστημα κλειδώματος αλκοολόκ που το λένε ε, ασφάλεια. Προσπαθήστε να πάρετε ασφάλεια ε, για το αυτοκίνητό σας αν έχετε υποπέσει σε αδίκημα ε, λόγω μέθης, ε, γιατί οδηγούσετε σε κατάσταση μέθης, θα καταλάβετε πώς μπορούμε με τις περιοριστικές ρυθμίσεις να εφαρμόσουμε την καλύτερη τέτοια ρύθμιση κλειδώματος κατά της οδήγησης υπομέθη. Οι όλοι, οι όλες αυτές οι προτάσεις λοιπόν ε, χρειάζονται αρκετά σχόλια. Έχω διδαχθεί και από τις τοπικές αρχές αυτοδιοίκησης στη δική μου χώρα και στη δική μου εκλογική περιφέρεια ότι υπάρχουν πάρα πολλά οδικά σήματα, τόσα πολλά που μπλέκουν και μπερδεύουν τους οδηγούς μάλλον παρά τους διευκολύνουν. Μιλάμε Μιλάτε επίσης στην έκθεσή σας για τη δημιουργία ενός συντονιστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο ένα γραφειοκράτη. Τι να τον κάνουμε. Θέλουμε περισσότερα, μεγαλύτερη συλλογή δεδομένων. Τι θα τα κάνουμε. Περισσότερη γραφειοκρατία και μεγαλύτερο κόστο και μάλιστα σε μια στιγμή που όλε οι κυβερνήσει, όλα τα κράτη προσπαθούν να μειώσουν τι δαπάνε του. Και εμεί εδώ λέμε ότι πρέπει να δαπανίσουμε περισσότερα χρήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και άλλο ένα σχόλιο έχω για τα FEE, e συστήματα περιορισμού ταχύτητα. Τι είναι αυτά τα συστήματα, εννοείται συστήματα περιορισμού τη ταχύτητα. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να ψηφίσω ε, υπέρ του να περιορίσουμε την ταχύτητα στα ιδιωτικά οχήματα, στα επιβατικά οχήματα. Αυτό είναι ε, θέμα που ε, κατά κανένα τρόπο δεν θα μπορέσουμε εμείς να, να το περάσουμε. Ούτε για συστήματα όπως τον Καλλιλέο μπορούμε εμείς να προτείνουμε να εφαρμοστούν. Νομίζω ότι είναι κρίμα που καταλήξαμε σε κάτι τέτοιο. Η κυρία Γκρίσπεκ νομίζω ότι είχε δίκιο όταν είπε ότι πρέπει να εξετάσουμε την ε, εφαρμογή διασυνοριακά. Η εφαρμογή σε διασυνοριακό επίπεδο μέχρι τώρα αφορά τα πλημελήματα. Ε, εγώ θα συμφωνούσα αν μιλούσαμε και για πιο σοβαρά αδικήματα. Προ το παρόν η αστυνομία θεωρεί ότι είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει τα πιο σοβαρά δικήματα διασυνοριακά και αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα δεν υφίστανται τις απαραίτητες κυρώσεις. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε λιγότερες περιοριστικές ρυθμίσεις, καλύτερη ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών και θα σας βοηθήσω κύριε Πρόεδρε ε, να μειωθεί η έκταση της έκθεσης του κυρίου Κόχ. Εγώ θα προτείνω να διαγραφούν πολλές παράγραφοι. Ευχαριστώ κύριε Μπράντμπορν. Ε, δεν με εκπλήξατε με αυτά που είπατε κύριε Ράνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο κύριο Κόχ για την έκθεσή του να συγκρατήσουμε αυτό το οποίο είναι πιο σημαντικό και ίσως ε, να παραλείψουμε αυτά τα οποία είναι λιγότερο σημαντικά. Θα συμφωνήσω για κάποια σημεία με τον προηγούμενο ομιλητή. Αυτός ο συντονιστής τι ακριβώς θα κάνει. Είναι αποτελεσματικό να έχουμε ένα τέτοιο συντονιστή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. ένα καθήκον ενός συντονιστού θα ήταν να βελτιώσει την οδική ασφάλεια, να συντονίζεται καλύτερα η οδική ασφάλεια με βάση μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την οδική ασφάλεια. Υπάρχουν ενδείξεις ε, για τα οδικά σήματα σε αυτοκινητοδρόμους ε, και ε, Υπάρχουν ε, δυνατότητες για πιο ομοιογενή σήματα, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για εναρμόνιση σε απόλυτο επίπεδο. Οι διατάξεις για τις οδικές μεταφορές και για την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη δεν είναι εναρμονισμένες και εδώ θα μπορούσε να υπάρξει κάποια βελτίωση. Υπάρχουν πολύ διαφορετικά πρότυπα ασφάλειας ε, τα οποία θα μπορούσαμε ε, να προσεγγίσουμε. Και θα μπορούσαμε επίσης ε, να βελτιώσουμε τον έλεγχο. Χωρίς έλεγχο σίγουρα δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τις σωστές αρχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κρατήσουμε από αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Μπάτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Κόχ για την έκθεσή του. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση προσπαθούμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε δύο στοιχεία τις διαφορές που υπάρχουν ε, ανάμεσα στα νομικά συστήματα των ε, κρατών μελών και εγώ το ξέρω αυτό γιατί χρειάζεται να περάσω από πολλά σύνορα χωρών μιας και προέρχομαι από μια μικρή χώρα και ξέρω ότι είναι δύσκολο να προσαρμοστεί κανείς σε όλα τα διαφορετικά συστήματα από τη μια χώρα στην άλλη. Δεν είναι λοιπόν τόσο απλό. Την κινητικότητα θέλουμε να την προωθήσουμε και ακριβώς επειδή πρέπει να βελτιώσουμε την κινητικότητα και παράλληλα να τηρήσουμε αυτά τα οποία χρειάζονται για την οδική ασφάλεια και για τους κανονισμούς, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται αυτή η δυνατότητα, αυτή η μεγάλη προσπάθεια. Όσον αφορά το Vision Zero, αυτή την προσπάθεια επίτευξης μηδενικού αριθμού θυμάτων, καταλαβαίνω αυτά τα οποία απαιτούνται ε, και υπάρχουν και επιμέρους στόχοι μείωση των ατυχημάτων κατά 60% ε, για τα παιδιά και κατά 40% ε, αν αρχίσουμε να συζητάμε με ποσοστά νομίζω ότι αυτό ήδη έρχεται σε αντίθεση με την πρωτοβουλία για μηδενικό αριθμό θυμάτων. Για αυτό που είπατε τώρα για τη διαβίου μάθηση, διαβίου εκπαίδευση, μπορεί ε, να ε, ε, είναι οι συνάδελφοι πολύ καλοί οδηγοί και να μην χρειάζονται νέα εκπαίδευση. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδεύουμε σωστά τους οδηγούς για να βελτιώνουμε την οδική ασφάλεια. Ο συνάδελφος Κοχ κάνει μια πρόταση και για ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο και για τη θέση ενός Ευρωπαίου συντονιστού για την οδική ασφάλεια. Νομίζω ότι θα χρειαστούμε κάποιο ευρωπαϊκό οργανισμό αργά ή γρήγορα για την οδική ασφάλεια ε, και ξέρω ότι υπάρχουν αντιφάσεις για το θέμα αυτό, αλλά αυτή είναι η δική μου προσωπική γνώμη. Ευχαριστώ κύριος Γκρός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Κοχ και θα είμαι σύντομος. Νομίζω ότι ήδη υπάρχουν διατάξεις που μπορούν να βελτιώσουν την ασφάλεια. Ε, τους, ε, παραδείγματος χάρη διατάξεις για το χρόνο οδήγησης και για το χρόνο ανάπτυξης, ε, για το χρόνο ανάπαυσης, συγγνώμη. Υπάρχουν ε, δηλαδή διατάξεις που έχουμε ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πρέπει να τηρήσουμε καλύτερα, να εφαρμόσουμε καλύτερα, να δούμε πώς γίνεται ο έλεγχος αυτών των διατάξεων και η εφαρμογή τους στην πράξη. Ένα δεύτερο θέμα είναι η έλεγχη. Κάθε περιφέρεια, κάθε κοινότητα, κάθε χώρα έχει τη δυνατότητα ελέγχων, γιατί χιλιάδες πινακίδες μπορούμε να βάλουμε. Αν δεν υπάρχει σωστός έλεγχος, δεν πρόκειται να μας προσφέρουν τίποτα οι νέες ταμπέλες και τα νέα σήματα. Χρειάζονται λοιπόν οι έλεγχοι, το έχουμε πει πολλές φορές. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερους ελέγχους και κατά τη διάρκεια των ελέγχων θα πρέπει να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν για εναρμόνιση των κυρώσεων. Θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα μετρήσεων. Ο συνάδελφος ε, μίλησε για τον αριθμό των ε, νεκρών. Δεν λέμε ότι θέλουμε να έχουμε 18.500 θέματα. Θέλουμε να έχουμε 18.500 λιγότερα θύματα. Και κάθε θύμα λιγότερο για μας ε, είναι σημαντικό. Φανταστείτε τι, τι γλιτώνουμε αν σκεφτείτε πόσα δαπανά η ιατρική για να γλιτώσουμε τη ζωή ενός και μόνο ασθενούς. Θα πρέπει να δείξουμε λοιπόν αποτελεσματικότητα και ενότητες αυτά τα οποία θέλουμε να επιτύχουμε. Και συμφωνώ με τον Φίλιπ Μπράντμπουλ σε ένα σημείο ότι η πολιτική δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ευθύνη των εμπλεκομένων. Ε, θα πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα την ανάληψη ευθύνης σε προσωπικό επίπεδο. Και εδώ παίζει ρόλο και το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο. Όταν ξέρουμε ότι η ταχύτητα, το αλκοόλ και οι υποδομές είναι τρεις βασικές αιτίες των σοβαρών ατυχημάτων και αν εμείς ως χώρα ή ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνουμε τίποτα για να μειώσουμε αυτές τις παραμέτρους κινδύνου δεν χρησιμεύει να κάνουμε συζητήσεις και να λέμε ότι οι άλλοι θα πρέπει να αλλάξουν. Αν έχουμε κάποιον ε, που κάθεται στο τιμόνι με τρία ε, της χιλής ε, αλκοολομετρία. Νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο να συζητάμε τίποτα παραπάνω. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να θεωρηθεί αθώος αν δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τέτοια θέματα. Ευχαριστώ κύριος Χίγινς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να συνάδω με αυτούς και κύριο για την εξαιρετική έκθεση Μερικά σημεία τα οποία στην παράγραφος 20 Ε, ότι θα πρέπει να υπάρχει κατάρτιση αυτή τη στιγμή από αυτά τα χήματα. Νομίζω πως αυτό που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να βελτιώσουμε την τεχνολογία. Ε, να μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια δυνατότητα να υπάρχει αντίδραση εκ μέρους του, ε, του οδηγού. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχουμε, αν πάτε αυτή τη στιγμή ε, στο ίντερνετ θα δείτε πραγματικά ότι η οδήγηση γίνεται ένα από τα μεγαλύτερα πρόβλημα με τα οποία υπάρχουν εκεί πέρα και νομίζω πως θα ρυθμιστεί. Δεύτερο, σε σχέση του κύριου Κρίσπερκ, συμφωνώ όσον αφορά τις κυρώσεις, την εναρμόνιση κλπ. για τα οποία μιλάει. Φίλοι, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υπάρχουν λιγότερες κυρώσεις. Εγώ έχω από ένα νησί το οποίο είναι αυτή τη στιγμή πάρα πολύ μικρό Πηγαίνουν όμως αυτοί από το νησί πηγαίνουν στην ε, υπηρετική το που λέγαμε η Ιρλανδία, η οποία ε, κάνουν εκεί τις δοκιμές και μετά έρχονται στο... Θα πρέπει λοιπόν η Φιλανδία, Σουηδία και εμείς θα πρέπει να έχουμε ένα έλεγχο όπου θα πάτε σε ένα οφθαλμίαρχο να υπάρχει μια γραπτή επιβεβαίωση αυτή τη στιγμή ότι μπορείτε να βλέπετε πολύ καλά και να επισυνάπτε και αυτό. Ο Φίλιπ Μπάμ τώρα έκανε μια παρατήρηση και θα πρέπει να επανέλθω σε αυτήν από το μετά το Μάστριχ όσον αφορά την ελεύθερη διακίνηση των υπηρεσιών, των κεφαλαίων και των ατόμων. Ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε μία ε και αν έχουμε μεταφορές οι οποίες, εκείνο το οποίο θα πρέπει να έχουμε όχι 27 διαφορετικά κανονισμούς αλλά πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση όσον αφορά και να ε, κάτι το οποίο ισχύει στην Α χώρα θα πρέπει να υπήρχε και στη Β χώρα εφόσον αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο συνάδει με την γενική ασφάλεια. Επίσης θα πρέπει για το θέμα της ταχύτητας να υπάρξει και εκεί μία εναρμόνιση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενος αγορητής παρακαλώ έχει το λόγο. Πρόεδρε ευχαριστώ. Μια εναρμονιση ευχαριστω παρα πολυ επόμενο αγορητης παρακαλω εχει σύντομη. Συγχαρτήρια και εγώ στον κύριο Κοκ για την εργασία του, την ιδιαίτερα λεπτομέρη. Να προσθέσω μόνο μια παρατήρηση. Ήδη Νάταλη Γκρισμπέγκ εξέθεσε την θέση της ομάδας μου και μάλιστα πολύ καλά. Η παρατήρησή μου τώρα. Πολλές πτυχές λαμβάνονται υπόψη σε αυτό. Τα θύματα, τι γίνεται σε αστικές ή μη αστικές περιοχές, η κυκλοφορία, όλα αυτά. Αλλά κάτι λείπει. Πολλά ατυχήματα πότε συμβαίνουν. Το Σαββατοκύριακο. Ίσως το στοιχείο αυτό να λευθεί υπόψη ώστε στις ρυθμίσεις τις εθνικές να ληφθούν υπόψη και τα ατυχήματα παθαίνουν κυρίως οι νέοι. Και δυστυχώς το σημείο αυτό δεν έχει συμπεριληφθεί στην ε, εξέταση του θέματος και στην αναπτυξή του. Ο συνάδελφος Μπράτμπορν ε, που είπε κάτι με έκανε να σκεφτώ και εγώ ότι ίσως ε, να προταθεί μια τροπολογία για να ρυθμιστούν τα πράγματα σε όλη την Ευρώπη. Γιατί άλλοι πάνε δεξιά, άλλοι πάνε αριστερά. Ίσως ο Μπράιν συμφωνήσει. Να πω το αστιάκι μου, έτσι. Ίσως η Μεγάλη Βρετανία έτσι να πάει λίγο πιο αριστερά. Αλλάζοντας λωρίδα κυκλοφορία. Εγώ πάντα έλεγα πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουν οι Βέλγοι, να οδηγούμε στη μέση του δρόμου ως συμβαστική λύση. Κυρία Σενιαλόβα. Eh, Πολλά ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση και έχω τρεις συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Ορισμένοι ομιλητές ανέφεραν την παράγραφο 20. Στην παράγραφο 20 μιλάμε για την εκπαίδευση των οδηγών και αναφέρονται και συγκεκριμένοι τομείς ε, όπως η χρήση ζώνη ασφαλείας ε, και προστατευτικού εξοπλισμού. Εδώ θα ήθελα να πω ότι παράλληλα με τα μέτρα αυτά καλό θα ήταν να υπάρχει καλύτερη εκπαίδευση ε, για την οδήγηση, γιατί υπάρχουν επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης το χειμώνα, παραδείγματο χάρη με τον παγετό ή το χιόνι και η ασφαλής οδήγηση θα έπρεπε να είναι τμήμα της ε, εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων οδηγών. Ακόμη, πιστεύω ότι η κοινωνία δεν πρέπει να ανέχετε επικίνδυνες συμπεριφορές στην οδήγηση. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να συνεργαστούν και οι πολίτες. Υπάρχει Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις ασφαλείς μεταφορές και θα πρέπει να συνεργαστούμε περισσότερο σε αυτό τον τομέα. Τρίτη παρατήρηση. Όταν μιλάμε για τις πιο ευάλωτες ομάδες των χρηστών, τους μοτοσυκλετιστές και τα παιδιά συγκεκριμένα, θα ήθελα να προσθέσω εγώ και τους ηλικιωμένους. Γιατί σαφώς και οι ηλικιωμένοι είναι ευάλωτη κατηγορία όσον αφορά τις οδικές μεταφορές. Κυρία Γιάλα. Με ναι, ευχαριστώ πρόεδρο. Συγγνώμη, καθυστέρησα γιατί ήμουν στον προπολογισμό και με την απαλλαγή είχαμε κάτι προβλήματα. Για τον κύριο Κόχ να τον ευχαριστήσω για την προσπάθεια του, την τεράστια για το θέμα αυτό και πάντα συνεργαζόμαστε όσο καλύτερα μπορούμε και συμφωνούμε με το ότι θα πρέπει να και τα ηλικιωμένα άτομα να συμπεριληφθούν και σαν ευαίσθητα άτομα, ευάλωτα και σαν ε, ενεργά άτομα για το τι έχει να κάνει με την υγεία και με διάφορες άλλες πτυχές μιας Ευρώπης που γερνάει όλο και περισσότερο και θα πρέπει να λάβει υπόψη της αυτές τις ομάδες τις ηλικιακέ. Και επίσης οτιδήποτε έχει να κάνει με τις ε, μοτοσικλέτες ε, και έχουμε πολλά θύματα, τώρα σε σύγκριση με τα αυτοκίνητα και από τους τουρίστες και ασκείται μια πολεμική δηλαδή δεν πρέπει να ξεχνάμε ε, τι γίνεται με τα φώτα τους, το, το άλλο είναι ευαίσθητα σημεία και ότι αυτοί οι χρήστες. Θα πρέπει να το δούμε λοιπόν και θα πρέπει να τους λάβουμε ιδιαίτερα υπόψη σε κάθε πτυχή και για τα όρια ταχύτητος. Βλέπω ότι και ο Σκόχ μιλάει σε εθνικό επίπεδο για όρια ταχύτητος και θα πρέπει να διατηρηθούν και να δούμε πώς θα εντάξουμε την κατάσταση στα πλαίσια επίσης τα ευρωπαϊκά, να δούμε τι γίνεται και με τα καύσιμα θα το δούμε και αυτό και θα ήθελα στο όλη θέμα να βάλω αυτούς τους ε, μηχανισμούς για περιορισμό ταχύτητας και να τα δούμε, να δούμε επίσης και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είναι το στίχημα το ευρωπαϊκό το σημαντικό, χρειάζεται να το αναφέρουμε και αυτό και ο κύριος Καχ Κόχ νομίζω ότι συμφωνεί με αυτή την τοποθέτηση και για την υποδομή να ελέγχουμε το τι γίνεται με τα οδικά σήματα. Είναι πολλά περίπλοκα μπερδεμένα. Γι' αυτό λοιπόν με τη σήμανση αυτή θα πρέπει να την προσέξουμε. Είναι σημαντικό βασικό σημείο και εντάξει να είναι και έξυπνα αυτά τα σήματα και από τη στιγμή που τα συνδυάζουμε με τα αυτοκίνητα και με το λιποδομή να δούμε να κάνουμε μια εκτίμηση της χρησιμότητας για να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα και δυσκολίες. Και ακόμα η οδική ασφάλεια στις πόλεις μέσα είναι κάτι που θα πρέπει να ενισχύσουμε στα πλαίσια αυτής της ευκαιρίας μας προσφέρεται. Ευχαριστούμε. Τέλος, θα ήθελα εγώ να πω λίγα λόγια. Θυμάμαι πάντοτε, κύριο Ζίασεν, ο κύριο Βιντάντσε έχει φύγει, ο κύριος Γκάντιαν επίσης, έβλεπα μεγάλη ε, γοητεία θα έλεγα με μεγάλο θαυμασμό αυτή τη στιγμή έναν Ιταλό αστυνομικό ο οποίος ότι πραγματικά βρισκόταν πάνω στο στο βήμα του και έδειχνε πραγματικά πώς θα πρέπει να, να, κυκλοφο... γίνεται η κυκλοφορία. Αυτό θα πρέπει να γίνει και στις Βρυξέλλες Αυτό το οποίο προσπαθώ εγώ αυτή τη στιγμή είναι να, κανονίσει, υπάρχει ο, ένας κανονισμός ο οποίος θα προβλέπει αυτή τη στιγμή τι θα πρέπει, ε, πώς θα πρέπει να οδηγούν οι οδηγοί. Υπάρχουν βεβαίω οι περισσότεροι που είναι καλύτερα, υπάρχουν και μερικοί που είναι φρικτοί αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να δούμε πραγματικά όταν ξεκινά 17 ή 18 χρόνια στην Ευρώπη και παίρνει την άδειά σου, κάνει πραγματικά ε, ε, τότε περάσει την έκθεση Κατά πόσο όμω τα 60 επόμενα χρόνια μπορεί να είσαι τέλειο, όχι δεν μπορεί να γίνει. Ξέρετε ότι σταδιακέ τα πραγματικά μειώνονται, διότι όσο γερνάει κανείς τα πράγματα επιδεινώνεται. Έτσι λοιπόν από τα 17, όταν περνάει ένα τεστ, όπου πραγματικά πηγαίνει με 50 miles μόνο, όταν ε, στα 75 πηγαίνει στο δρόμο με 15 μόνο miles έτσι λοιπόν αυτό είναι ο λίγο. Ε, μπορείτε να το προκαλέσετε αυτό όπω θέλετε εσεί και να δείτε πραγματικά όλου του δρόμου που έχουν. Αλλά θα πρέπει να δούμε όταν εξετάζουμε αυτό το θέμα ότι είναι πολιτικά απαράδεκτο αυτή τη στιγμή να επιτιθέμαστε εναντίον των οδηγών. Όλοι οι πολιτικοί οι οποίοι πραγματικά φοβούνται να τα βάλουμε τους οδηγούς αυτοκίνητα αλλά θα πρέπει να το κάνουμε αυτό το στιγμή διότι οι ιδιώτες είναι φρικτοί πραγματικά είναι εντελώς κυκλοθυμική μερικές φορές για αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να δούμε πραγματικά, μπορούμε να πούμε ότι στα 17 χρόνια κανείς ο οποίος ξεκινάει ε, μπορεί να φτάσει αυτό το τέλος του πεζίτη. Πώς μπορεί αυτό πραγματικά κατά πόσο πραγματικά τον αφήνει σε μια προκεχωρημένη ηλικία ή αν δεν έχει πάρει την άδεια, τον αφήνει στον δρόμο ξε, ατέσποτο για να σκοτώσει τον κόσμο. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Θα πρέπει να μιλάμε βεβαίω για τα δικαιώματα του οδηγού, αλλά πού είναι τα δικαιώματα των θυμάτων τα οποία υποφέρουν αυτό το θέμα. Ξέρετε, έχασα ε, ένα συγγενή ακριβώς γιατί κάποιος μιλούσε στο κινητό ενώ οδηγούσε. Καταλαβαίνετε τι γίνεται λοιπόν. Θα πρέπει να το δούμε λοιπόν του αυτό. Ανεφέρθηκε επίση θέματα όσον αφορά την τεχνολογία. Εάν πραγματικά δεν είσαι σε θέση, δεν θα πρέπει να παίρνει μπροστά η μίζα. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύω θα πρέπει να σταματάει το πράγμα, γιατί θα πρέπει να το κάνουμε, γιατί ξέρετε ε, ότι μερικοί βάζουν στον νεκρό, ξεκινάνε και μετά. Είναι αυτά θέματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε για να αποφύγουμε αυτή τη φρικτή κατάσταση οποία... Όσον αφορά την εφαρμογή τη διασυνοριακή, πιστεύω σε αυτό το οποίο είπες προηγουμένως Φίλιππ, στο Ηνωμένο Βασίλεια, κοίταξε τι έγινε αυτή την εβδομάδα, γιατί θα πρέπει να υπάρχει δεν πρέπει να είναι αναποφάσιστα. Θα πρέπει να υπάρχει, να τεθεί το θέμα και να αποφασιστεί. Επίσης, όταν δείτε τις υπηρεσίες οδικής βοήθειας θα πρέπει πρέπει να δείτε πραγματικά τι είναι το Βασίλειο πριν οδηγήσετε εκεί πέρα τι γίνεται. Γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες λακκούβες, υπάρχουν τόσο, τόσα προβλήματα και υπάρχουν τόσες συγκρούσεις οι οποίες Νομίζω πως πραγματικά η οδική βοηθήθεια είναι το πιο βασικό πράγμα το οποίο μπορεί να υπάρχει. Πριν κανένας λοιπόν αυτή τη στιγμή φτάσει σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένοι οι δρόμοι για να μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν υπάρχει κακό υποδομή, υπάρχουν τα φορτηγά, υπάρχουν πολλά ατυχήματα και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο εκεί είναι τα προβλήματα, εκεί είναι τα κενά τα οποία υπάρχουν. Και οποιοδήποτε κάνει αυτό το πράγμα θα πρέπει να σταματήσει να το κάνει αυτό εγώ με αυτό το δρόμο δεν γίνομαι εναντίον τη ε, οδική φραγματέτηση ούτε εναντίον τη επιχείρηση, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα, γι' αυτό ήθελα να το καταθέσω. Ε, εκ μέρου τη εκμετροπή ο εκπρόσωπο, παρακαλώ. Δεν ξέρω τι να πω. Καταρχήν να σα ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κύριο Κόχ για την εξαιρετική του έκθεση και για την υποστήριξή του προς την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κατευθυντήριε γραμμές 2011-2020. Η Επιτροπή χαίρεται διότι βλέπει ότι οι τρει πυλώνες, δηλαδή επιμεριζόμενη ευθύνη, η ολοκλήρωση και οι κανόνες οδικής ασφάλειας συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση. Όσον αφορά την επιμεριζόμενη ευθύνη, η Επιτροπή χαίρεται διότι ο εισηγητής δεν ζητάει μόνο από την Επιτροπή να αναλάβει δράση, αλλά και από τα κράτη-μέλη και από τη βιομηχανία. Ακόμη ο εισηγητής ε, υπενθυμίζει ότι οι πολίτες βρίσκονται στην καρδιά της οδικής ασφάλειας και συμφωνούμε απολύτως. Και η επιτυχία οποιασδήποτε πολιτικής οδικής ασφάλειας εξαρτάται από τη συμπεριφορά όλων των χρηστών του οδικού δικτύου. Δεύτερον, συμφωνώ με τον εισηγητή ότι η ολοκλήρωση, η ένταξη της οδικής ασφάλειας σε άλλες πολιτικές είναι το κλειδί της επιτυχίας. Η οδική ασφάλεια είναι βασική βασική παράμετρος και για την δημόσια υγεία και για και άλλοι τομείς όπως η αλλαγή του κλίματος ε, έχουν άμεση ε, σχέση και ε, η τεχνολογία και τα ηλεκτρικά οχήματα. Οι βέλτιστες πρακτικές και οι κατευθυντήρες γραμμές θα είναι απαραίτητες καθώς και η διάδοσή τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τώρα, να κάνω ορισμένα σχόλια στις προτάσεις που κάνει η έκθεση. Όλοι συνεργαζόμαστε προς το μηδενικό αριθμό θυμάτων, αλλά θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω στο πρόγραμμα δράσης οδικής ασφάλειας ε, με τον οδικό χάρτη που προτείνουμε και θα λάβουμε υπόψη και τις δικές σας συστάσεις. Δεύτερον, για την πρότασή σας για το συντονιστή οδικής ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα συμφωνήσω με κάποιους ομιλητές που είπαν ότι πρέπει πρώτα να ορίσουμε το ρόλο που θα παίξει ένα τέτοιο συντονιστή. Πάντως η Επιτροπή θα εξετάσει την πρότασή σας κύριε Σιγητά για την μείωση του αριθμού των πόν που είναι θύματα κατά 60% και για τη μείωση άλλων κατηγοριών συγκεκριμένων κατά 40%, νομίζω ότι είναι δύσκολο να βάλουμε συγκεκριμένους στόχους και είπε και κάποιος άλλος ομιλητής ότι αν βάλουμε τέτοιους στόχους μείωσης, αυτό είναι αντιφατικό προς, την, προς το όραμα του μηδενικού αριθμού θυμάτων. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές και το συντονισμό των πολιτικών μας. Τέλος, στην εναρμόνιση των οδικών σημάτων και των κωδίκων οδική κυκλοφορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν θετικά στοιχεία. Γνωρίζετε όμω ότι όπω και στην εναρμόνιση των ορίων ταχύτητα μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο να καταλήξουμε σε συνένεση μεταξύ των κρατών μελών. Η εναρμόνιση των οδικών σημάτων είναι επίσης ένα θέμα το οποίο αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων σε πολυεθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της UNICEF, παραδείγματο χάρη. Είμαστε πεπισμένοι ότι σε συνεργασία θα επιτύχουμε καλύτερη οδική ασφάλεια για τους πολίτες της Ευρώπης στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής μέχρι το 2020. Ευχαριστώ πολύ και πάλι τον κύριο Σίγητη. Ντίτα, θέλεις να λάβεις το λόγο κλείνοντας αυτή τη συζήτηση. Μου δίνετε μία ώρα, πόση ώρα μου δίνετε. Δέκα λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Ελκαντράουι και άλλοι μίλησαν για το θέμα του συντονιστού και το επανέλαβε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπα στην παρέμβασή μου ότι το θέμα της οδικής ασφάλειας είναι κάτι το οποίο ε, θα πρέπει να αντανακλάται σε όλους τους τομείς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και στη γεωργία και στον πολιτισμό και στο περιβάλλον παντού. Και αυτός ο συντονισμός λοιπόν είναι απαραίτητος και γι' αυτό χρειάζεται ένα συντονιστή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ότι ε, θα πρέπει αυτός ο συντονιστής να λάβει υπόψη και ε, τα εθνικά προγράμματα δικής ασφάλειας των κρατών μελών. Ελπίζω να μπορέσει να δημιουργηθεί μια τέτοια θέση συντονιστού. Προς τον κύριο Ελκαντραουή θέλουμε να έχουμε συγκρισιμότητα και συμφωνώ απολύτως ε, γιατί δεν έχω πει παιδιά μέχρι την ηλικία των 14 ετών γιατί νομίζω ότι από αυτή την ηλικία και πάνω τα παιδιά αρχίζουν να, μαθαίνουν περισσότερο τα, θέματα της οδικής ασφάλειας και ε, σιγά σιγά αρχίζουν να παίρνουν και δίπλωμα. Επομένως μέχρι την ηλικία των 14 ετών είναι η πιο επικίνδυνη ηλικία. είπε ο κύριος Μπράτμουν ότι δεν χρειάζεται κατάρτιση. Να σας βάλω εγώ 10 ερωτήσεις και θα δείτε ότι σε μερικές από αυτές τις ερωτήσεις μόνο κατά τύχη θα απαντήσετε σωστά. Είπατε ότι έχετε δεν ξέρω πόσα χρόνια, είπατε 40 χρόνια δίπλωμα οδήγηση και μαθαίνετε κάθε μέρα. Μα δεν το πιστεύω ότι κάθε μέρα μαθαίνουμε και δεν χρειαζόμαστε περαιτέρω εκπαίδευση. Για τη διαμεθοριακή τώρα ε, επιβολή των διατάξεων Υπάρχουν πολλές δυσκολίες στην επιβολή διασυνοριακά. Για την εναρμόνιση των οδικών σημάτων και των πινακίδων, θα πρέπει να είναι πληροφορίες ε, που να είναι πιο εύκολα κατανοητές. και μια εφαρμογή του συστήματος πλοήγηση μέσω του Γκαλιλαίου είναι επίση κάτι το οποίο μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας. Μέχρι το 2020 το Vision Zero, ο μηδενικό αριθμό θυμάτων, δεν είναι εφικτό. Ε, είπα ότι θέλουμε να έχουμε εφικτού στόχου και γι' αυτό είπα ότι το όραμα του μηδενικού αριθμού θυμάτων ε, πρέπει να το έχουμε κατά νου σαν απότερο στόχο. Πιο μακροπρόθεσμα και όχι μέχρι το 2020. Νομίζω ότι μπορούμε να προσβλέπουμε στον, στη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων, αλλά όχι μηδενικό αριθμό μέχρι το 2020, γιατί δεν το θεωρώ εφικτό αυτό. Το να έχουμε εναρμόνιση κάποιων ε, νομικών πλαισίων ε, είναι όντως ε, κάτι χρήσιμο. Ε, αυτό που ο κύριος Γκρός για την ευθύνη που έχει ο καθένας από εμά και βέβαια είναι πολύ σημαντικό ε, όλοι εμείς που συμμετέχουμε στις οδικές μεταφορές υπό οποιαδήποτε ιδιότητα φέρουμε ευθύνη και θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ούτω ώστε να υπάρξει πλήρης επίγνωση όλων. Γιατί όλοι γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας και θέλουμε να έχουμε δικαιώματα αλλά τα καθήκοντά μας και τα καθήκοντα που έχουμε στις οδικές μεταφορές δεν τα λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη μας. Νομίζω ότι χρειάζεται καλύτερη επίγνωση ε, του ότι ε, δεν μπορούμε να οδηγούμε υπομέθη, ε, πρέπει να φοράμε την ζώνη ασφαλείας κλπ. Νομίζω ότι η επίγνωση λοιπόν των υποχρεώσεών μας είναι πολύ σημαντικό θέμα. Προς την κυρία Γιάλα νομίζω ότι είναι λογική η πρότασή σας το είχαμε αναφέρει στην συντομία, αλλά δεν ήσασταν εδώ την ώρα που το είπα. Ευχαριστώ πολύ πάντως για την πρότασή σας, την οποία θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω. Εναρμόνιση των φωτεινών σηματοδοτών Ε, υπάρχουν έννοιες οι οποίες είναι παρόμοιες, αλλά ακολουθούνται διαφορετικές ρυθμίσεις στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν διαβάσεις πεζών με ή χωρίς φωτεινούς συμμετοδότες, παραδείγματο χάρη. Εδώ θα μπορούσαμε να εξετάσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν. Κύριε Σίμψον, ναι, και για τους μοτοσυκλετιστές έχετε δίκιο και για την συντήρηση του οδικού δικτύου. Βεβαίως έχετε δίκιο ότι έχει σημασία το οδόστρωμα και όταν υπάρχουν προβλήματα στο οδόστρωμα μετά από το χειμώνα, παραδείγματο χάρη στη Γερμανία, βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλε ζημίε λόγω των καιρικών συνθήκων το χειμώνα. Και χρειάζεται πολύ συχνά να μπουν πινακίδε που θα λένε ότι πρέπει να μειωθεί η ταχύτητα γιατί το οδόστρωμα έχει βλάβες. και συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να επιτηρούμε τους δρόμους ώστε να υπάρχει σωστή ποιότητα του οδικού δικτύου. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κόλλο. 14 Μαρτίου είναι η 14 ε, Μαρτίου λοιπόν είναι η προθεσμία όσον αφορά τις τροπολογίες και θα πάμε βεβαίω στην Ολομέλεια του Ιουνίου. Βεβάσια, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τους πάντες για την παρουσία τους και τη συμβολή και θα ξεκινήσουμε σε πέντε λεπτά του συντονιστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.